Να πω άλλη μια φορά ότι οι συνεδριάσεις μας μεταδίδονται στο διαδίκτυο και πριν περάσω στην ημερήσια διάταξη αυτή αυτή θα ήθελα να ζητήσω κάποιες αλλαγές. Τα σημεία 4 και 5 να μεταφερθούν στο σημείο 9, αν δεν σας πειράζει. Τότε αν δεν έχετε αντιρρήσεις, εγκρίνεται όσο έχει η ημερήσια διάταξη. Το πιλωτικό πρόγραμμα για τις ε, συνεδριάσεις χωρίς έγγραφα, δηλαδή τα έγγραφα να είναι διαθέσιμα μόνο ηλεκτρονικός, είναι ήδη πραγματικότητα. Αυτό είναι κάτι για το οποίο ενημερώνονται τα μέλη της Επιτροπής από τη Γραμματεία. Πρώτον, λοιπόν, Επιβεβαιώνουμε λοιπόν την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Και να δώσω το λόγο στον κύριο Ρότιν που δεν είναι εδώ όμως. Υπάρχει κανένας άλλος που να μπορεί εδώ να τον αντικαταστήσει. κολέγα ε, Δίνω το λόγο στον συνάδελφο Σφάμπ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ρόιτεβα δεν θα μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Όμως, μας είπε σε γενικές γραμμές τι την ενδιαφέρει ως προς την εναρμόνιση. Όσον αφορά λοιπόν την έκθεσή της, η έκθεση της κυρίας Ρόιτοβα και η συνέχιση της, ε, του πακέτου της ε, δέκατης ε, οδηγίας επί, την οποία, επί της έχει ήδη εργαστεί. Όλα αυτά είναι τμήμα των τμήματων, ε, είναι, τμήμα, είναι τμήμα της νομοθεσίας ε, που έχει να κάνει με τα εμπορεύματα. Υπήρξαν όμως ε, κάποιες αλλαγές για να υπάρξει συνεχή με τους υπόλοιπους με, τις με την υπόλοιπη νομοθεσία σχετικά με το θέμα αυτό. 15 Νοεμβρίου θα κάνουμε την τελική μας ψηφοφορία αν έχει ολοκληρώσει η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων τις δικές της εργασίες εγκαίρως. Δεν ξέρω όμως εάν η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων δεν θα αν θα προλάβει να ολοκληρώσει τις εργασίες της ως τότε. 53 τροπολογίες έχουν ε, κατατεθεί και η κυρία Ρόιτοβα προσπάθησε να υπάρχουν ε, λιγότερα εμπόδια για τους ε, καταναλωτές, ώστε να υπάρχει ένα αυστηρό πλαίσιο για την προστασία των καταναλωτών. Η κυρία Ρόιτοβα θα ήθελε να ευχαριστήσει τους συμβούλους και τους κοιόδης εισηγητέ. Είναι ανοιχτή σε κάθε σχόλιο. Δεν ξέρω κύριε Πρόεδρε αν θέλετε να σας διαβάσω συγκεκριμένες ε, αλλαγές που θα ήθελε να εισαγάγει η κυρία Ρόιτοβα. Έχω 11 σημεία τα οποία θα μπορούσα να σας παρουσιάσω αν θέλετε. Στα αγγλικά. Λοιπόν, πρώτον, η κυρία Ρόιτεβα θα ήθελε να αναφέρει νέα προϊόντα, δηλαδή να καλύπτουν και τα δεύτερο χέρι προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες. Ε, είναι κάτι το οποίο όμως το έχουμε κάνει στο πακέτο των υπολείπων εννέα οδηγιών, οπότε δεν είναι κάτι το πολύ καινούριο. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σας το πω. Δεύτερον, θα ισχύει για ε, όλες τις μορφές πωλήσεων ε, και για τις ηλεκτρονικές πωλήσει. Δεν θα καλύπτεται μόνο η ασφάλεια των, ανθρώπων, αλλά και η ασφάλεια ε, και μία άμεσα συνδεδεμένη περιουσία. Τέταρτον, θα γίνει μία αποσαφήνιση σε σχέση με τις, τα, τα στοιχεία με τα οποία μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με τους ε, κατασκευαστές. Θα υπάρχει μία ενιαία δήλωση συμβατότητας ε, που θα βελτιώσει την γραφειοκρατία. Και έβδομον, αποσαφηνίζεται ότι η οδηγία καλύπτει όχι μόνο τα, τον εξοπλισμό υποπίεση αυτό καθ' αυτόν, αλλά και τα άλλα εξαρτήματά τους. Και αυτό είναι το τελευταίο που θα ήθελα να πω κύριε Πρόεδρε. θα, θα μπορούμε να, να επιβάλλουμε περισσότερες κυρώσεις σε περίπτωση που δεν είναι καλή η εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Ελπίζω ότι έλαβα υπόψη είναι παρκώς επιθυμίε τη κυρίας Ρόιτοβα για να σας παρουσιάσω τη διαδικασία και ελπίζω να μην εξαντλήσα την ε, υπομονή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Collega, e, passiamo al Μάλιστα. Πολύ ωραία, συνεχίζουμε. Πάμε τώρα στους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβιάση των διατάξεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Φαμπ ε, είναι ο επί της ουσίας ε, εισηγητής για την Επιτροπή Οικονομικών. Δίνω το λόγο όμως για την ώρα στον κύριο Σμιτ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είναι γεγονός ε, ότι ο κύριος Φάμπ είναι ο πιο αρμόδιος και χαίρομαι που είναι εδώ. Είναι πολύ καλό για όλους μας αυτό. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό το ότι ο συγκητής μας είναι ο Ανδρέας ε, Σφάμπ. Ξέρετε ότι το δίκαιο του ανταγωνισμού ε, και από τις αρμόδιες αρχές επιβάλλεται, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία οι πρακτικές κατά του ανταγωνισμού είναι πολύ επιβλαβείς για την ευρωπαϊκή οικονομία και επηρεάζουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Μόνο μερικά κράτη-μέλη για την ώρα δίνουν τη δυνατότητα αγωγών και ε- αίτησης ε, ε, αποζημίωσης και αυτό σημαίνει ότι πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους. Νομίζω ότι πολλοί εξημών ε, χαιρετίζουν συνεπώς την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όσον αφορά τώρα την ιδιωτική επιβολή, εγώ έκανα το εξή. Ε, είναι καλό να συμπεριληφθεί η συλλογική αγωγή για αποζημίωση. Ελπίζω ότι ο κύριος Φαμπ μπορεί να, μας, να με ακολουθήσει σε αυτή μου την προσπάθεια γιατί έχει γίνει και ψήφισμα της, ε, του Κοινοβουλίου το 2009 που λέει ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τις συλλογικέ αγωγές, ε, για την αποκατάσταση και την αποζημίωση στο πλαίσιο του, του δικαίου ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρουμε βέβαια ότι κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει πραγματικότητα ακόμα, παρόλα αυτά, που, ε, παρόλα αυτά εγώ πάντοτε υπερψήφιζα κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε εσωτερική αγορά χωρίς ένα τέτοιο είδους μέτρο αλλά η συλλογική αποζημίωση θα δώσει τη δυνατότητα ε, εμπορικές ενώσεις, ενώσεις καταναλωτών ε, να υποβάλουν αγωγές εκ μέρους ε, του μεμονωμένου ενάγοντος θέλουμε να υπάρχει ένα θεματολόγιο καταναλωτή δίκαιο και πλήρες. Ζητώ απλώς μία σαφώς αναγνωρισμένη ομάδα ατόμων που θα μπορούν να δρουν ως αντιπρόσωποι ε, και να συμμετέχουν στην αγωγή. Ξεκινώ κάπως ε, γενικά, αλλά ξέρετε ότι η πολιτική πραγματικότητα στο τέλος πάντοτε υφίσταται. Πρέπει όλα αυτά να έχουν ολοκληρωθεί. Αυτή τη στιγμή αρχίζει η αγωγή και ελπίζω να υπάρχει ένα μοντέλο opt-in γιατί σε πολύ, σε πολύ λιγότερες περιπτώσεις ε, καταλήγουμε όντως σε αγωγή. Πρέπει περισσότεροι καταναλωτές να ενθαρρυνθούν, ε, να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και υποθέτω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Όσον αφορά τώρα ε, το, την... Ε, προσπάθεια μιας πιο ήπιας επίλυσης διαφορών. Δεν συμφωνώ ότι θα έπρεπε να ε, να ε, παρακρατώνται κάποια στοιχεία μέχρι να ολοκληρωθεί όλη η ε, αγωγή. Νομίζω ότι οι κανόνες της πρώτης παραγράφου του άρθρου 6 θα πρέπει να ισχύει ανεξαρτήτως αν ισχύει η αίτηση επίοικιας ή αν έχει γίνει αξιολόγηση της αίτησης από τις αρμόδιες αρχές. Σε μερικές περιπτώσεις ε, ε, πολλές, σε πολλές περιπτώσεις ε, υπήρξαν πληροφοριοδότες και γι' αυτό βρίσκω ότι δεν υπάρχει καμία ευελιξία ούτε λεπτομέρειες στην συγκεκριμένη πρόταση. Νομίζω ότι περισσότερα στοιχεία θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην πρόταση. Νομίζω ότι έτσι θα υπάρξει πραγματικά μία, ένα όφελος για τους άμεσους αγοραστές. Υπάρχουν όμως και οι έμεσες αγορές και δεν θα έπρεπε να υπάρχει ε, μόνο ε, το τεκμήριο. Αυτό σημαίνει ε, και άμεση και έμεση ενάγοντες. Εγώ πιστεύω ότι το σύστημα που προτείνεται δεν είναι επαρκές δεν είναι επαρκές για τη μετάβαση του άχθους της αποδείξεως, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα πυλώνων που να δίνει σαφείς οδηγίες στα εθνικά ε, δικαστήρια. Πρέπει κάθε, ε, κάθε ε, ζημία να αποζημιώνεται. Είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι όσοι προβαίνουν σε συλλογικέ αγωγέ ε, να έχουν τη δυνατότητα να την κερδίσουν ενώπιον του δικαστηρίου. Επίσης, αυτό ενισχύει τη συμμετοχή των ε, ε, Αυτό σημαίνει ότι σε μικρότερες ε, εταιρείε, μικρότερες επιχειρήσεις ε, θα πρέπει να πληρώσουν τεράστιες αποζημιώσεις και αυτό μπορεί να ε, δημιουργεί πρόβλημα στη δυνατότητα υποβολής αγωγών, κατάθεσης αγωγών. Γι' αυτό προτείνουμε θα μπορούσε σε αυτές τις περιπτώσεις να υπάρχει μια διαδικασία επιπαραβάση. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι θα υπήρχαν λιγότερες αγωγές και θα μειώνονταν ε, οι ε, μη απαραίτητες αγωγές. Παρ' όλα αυτά, ε, συμπερασματικά θα ήθελα να πω ότι επαφίεμαι σε αυτά που λέει ο κύριος Σφαμπ, του έχω πλήρη εμπιστοσύνη Είμαι σίγουρος ε, ότι θα τα καταφέρει πολύ καλά. Είμαι και εγώ πλήρες μέλος της ε, Επιτροπής Οικονομικών, οπότε ε, μπορώ βεβαίως να, σας, να σε υποστηρίξω εκεί, Ανδρέας, μπορεί και εσύ να με υποστηρίξεις εδώ. Θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες, αλλά για την ώρα αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ. <coughs> Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στον κύριο Σφάμπ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Όλε Σμιτ ε, με την ιδιαίτερη γοητεία του τα είπε όλα. Του, κάνω, του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Είμαι σίγουρος ότι αυτά που θα γραφτούν στην ε, γνωμοδότηση θα βοηθήσουν πάρα πολύ τους καταναλωτές, γιατί στην καθημερινή ζωή πολλοί ε, πολίτες μας είναι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις, όπως και οι καταναλωτές, πληρώνουν πάρα πολύ ψηλό τίμημα για τέτοιου είδους ε, αγωγές. Οπότε Νομίζω ότι θα βελτιωθεί πολύ η κατάσταση. Κάποιους από τους μηχανισμούς που έχουμε ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν, ε, έδωσαν τη δυνατότητα κάποιων αποζημιώσεων. Ελπίζω να συνεχίσει και να βελτιωθεί αυτό στο μέλλον. Γι' αυτό θα έπρεπε να αναρωτηθούμε κατά πόσο η Επιτροπή θα έπρεπε να ενισχύσει ενδεχομένως ε, το προσωπικό της για να μπορεί να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα ε, προβλήματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας μην το πάω ως εκεί για την ώρα. Θα ήθελα να σας μιλήσω για μία διάσκεψη. Ο Φιλίπ Κουμπίκ, ε, εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, είναι και εκείνο παρόν ε, και ο Όλε Σμιτ. Δεν θέλουμε δυσανάλωσιες αποζημιώσεις όπως γίνεται στις Ηνωμένε Πολιτείες, αλλά δεν θέλουμε δηλαδή να εισαγάγουμε το αμερικανικό μοντέλο, αυτό είναι σαφές, αλλά σε σχέση με το ερώτημα που ανέφερα εν είδη εισαγωγής, ε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια πραγματική ενιαία αγορά με κοινούς κανόνες. Ένας Ιρλανδός δικαστής ε, με, μου ερώτησε τι είναι το purity of damages στην Ιρλανδία. Κάτι το οποίο δείχνει ότι είναι διαφορετικέ οι παραδόσει για τι αποζημιώσει στα διάφορα κράτη-μέλη τη Ένωση και επομένω δεν θα μπορέσουμε να τα εναρμονίσουμε όλα όσον αφορά τι συλλογικέ αγωγέ. Είναι γεγονό ότι υπάρχουν ε, κάποιες, ε, ε, κάποια, κάποιες αποζημιώσεις, οποίες δεν θα μπορέσουμε να τις εναρμονίσουμε Όσον αφορά τώρα τα μεμονωμένα στοιχεία που ανέφερε ο κύριος Σμιτ, αν υπάρχει δηλαδή κίνδυνος να πέσουμε στην παγίδα, δεν νομίζω ότι δεν μπορούμε να προσπαθήσουμε οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, ή των ενώσεων καταναλωτών ε, ζητούν αποζημίωση, να μην αποζημιώνονται αυτοί οι άνθρωποι να εισακούγονται τουλάχιστον, τουλάχιστον. Γι' αυτό ακριβώς η άποψή μου είναι, και το έχω πει και στο παρελθόν, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως το δυνατόν περισσότερη εξουσία να αρχίσει μια διαδικασία, να βρίσκεται σε μια αρκετά άνετη θέση για να μπορεί να επιβάλλει ένα πρόστιμο σε, στο, στο ε, μέρος που έχει ε, προβεί ε, στην απάτη. Νομίζω ότι η προστασία των ε, μαρτύρων θα ήταν κάτι θετικό, αλλά στα άρθρα 5 και 6 καλύψαμε κάποια στοιχεία για να εξηγήσουμε ποια έγγραφα σημαίνουν ε, ευνοϊκή ε, πρόσβαση για όσους έχουν πληγεί από ένα καρτέλ. Είναι στοιχεία τα οποία ενδεχομένως πρέπει να τα επιβεβαιώσουμε πώς ε, η προστασία μαρτύρων θα έχει ως αποτέλεσμα να προστατεύονται τα δεδομένα τους, όχι μόνο του απορρίτου, αλλά και γιατί μας λείπει η εμπειρία. Όσο καλύτερα τα δεδομένα αυτά ε, κρατούνται, τόσο ε, λιγότερες καταχρήσεις θα υπάρχουν. Και νομίζω ότι μόνο έτσι θα επωφεληθούν πλήρως οι καταναλωτές. Κάποιοι μάρτυρες λοιπόν πρέπει να προστατεύονται αν αυτό συνάδει με τους εθνικούς κανόνες. Το ερώτημα τώρα του κυρίου Σμιτ θα πρέπει να υπάρχει μία μαύρη λίστα. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα να έχουμε μια γενικότερη θεώρηση και στη συνέχεια να δούμε κατά ποια, σε, ποιο βαθμό ε, θα έπρεπε τα στοιχεία αυτά να ε, τίθενται στη διάθεση ε, του ενάγοντος. Αλλά αυτά είναι στοιχεία που αφορούν μόνο την, την δικαστική διαδικασία. Για παράδειγμα, σε μερικές περιπτώσεις οι δίκες γίνονται σε διοικητικά δικαστήρια και μήπως θα έπρεπε να προβλέψουμε ειδικού κανόνες εν προκειμένου. Κάτι ακόμη που είπε ο κύριος Σμιτ. σε σχέση με την εθελοντική βάση της αποζημίωσης. Νομίζω ότι είναι η γρηγορότερη και η καλύτερη λύση, αλλά πρέπει πρώτα να μπορέσουμε να ασκήσουμε την πολιτική πίεση, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ε, όσοι έχουν υποστεί ε, τη ζημιά ε, θα αποζημιωθούν όσον αφορά τους έμεσους αγοραστές. Αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης πρέπει να το εξετάσουμε. Η αποζημίωση πρέπει να δίδεται μόνο στο επίπεδο της ζημίας και δεν θα έπρεπε ο αγοραστής, ο έμεσος, να μπορεί να χρησιμοποιεί την αποζημίωση αυτή. Γι' αυτό πρέπει πάρα πολύ σαφώς ε, να ορίσουμε την ιεραρχία των εναγόντων και να δούμε ποιο είναι το επίπεδο στο οποίο έχει γίνει μεγαλύτερη ζημιά, ώστε να μπορεί αυτό το, σε αυτό το επίπεδο να ασκηθεί ε, το σχετικό δικαίωμα. Δεν θέλω να πω βέβαια ότι σε κάθε περίπτωση ο ενάγων είναι αυτός που πρέπει πάντοτε να φέρει το βάρος αποδείξεως, αλλά τουλάχιστον πρέπει να μπορεί να γίνει μια αξιολόγηση Νομίζω όμως ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί δεν θα έπρεπε να είμαστε υπερβολικοί στο πόσο θα ενθαρρύνουμε κάτι τέτοιο. Πιστεύω όμως ότι θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.

Θα ήθελα να μιλήσω εκ μέρου τη κυρία Ράπτη, η οποία δυστυχώ ε, έχει ανηλυμένε υποχρεώσει στην Αθήνα και δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Θα ήθελα όμω ε, να σα διαβάσω το κείμενό τη ε, στα αγγλικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τον εισηγητή, τον κύριο Σμιτ, για την πολύ καλή ε, γνωμοδότησή του. Η πρόταση για την εν λόγω οδηγία είναι ένα ε, σημαντικό βήμα προς τα εμπρός που αναμενόταν και είχε ζητηθεί εντόνως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πολλά χρόνια παρά το ε, γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήταν αρκετά τολμηρή σε σχέση με την ε, συλλογική αποζημίωση των καταναλωτών, ε, εμείς χαιρετίζουμε αυτήν την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως πρώτο βήμα. Χαιρόμαστε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε σε δεσμευτικό νομικό πλαίσιο για να ορίσει και να εραμονήσει την ιδιωτική επιβολή σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα του ανταγωνισμού. Σε γενικές γραμμές η πρόταση καταδεικνύει πολλές ε, πολλά θετικά, πολλά ισχυρά σημεία. Αναγνωρίζει το δεσμευτικό χαρακτήρα των τελικών εθνικών αρχών ανταγωνισμού και των αποφάσεων των, αποφάσεων των τελικών των αρμοδίων αυτών αρχών. Ε, εξασφαλίζει το δικαίωμα του θύματος ε, σε αποτελεσματική αποζημίωση, όπως επίσης ε, και στη διευκόλυνση των συνενετικών ε, μηχανισμών επίλυσης. Επίσης, προσπαθεί να δημιουργήσει κοινέ αρχές για τους κανόνες πρόσβασης και της αποκάλυψης των αποδεκτικών στοιχείων. Ο καταναλωτής έτσι μπορεί να βρει πιο εύκολα τις πληροφορίες. Επίσης, επίσης ε, ε, ρυθμίζει την ε, και προστατεύει τη θέση των έμεσων αγοραστών, ενισχύει έτσι τους καταναλωτές και αντιμετωπίζει κάποιες ασυμμετρίες πληροφόρησης με σωστή εξισορρόπηση του βάρους της απόδειξης. Ο ενισχυμένος ρόλος των εθνικών δικαστηρίων στην αξιολόγηση ε, το, της αποζημίωσης ε, υπό την ε, ε καθοδήγηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής πηγαίνει προς σωστή κατεύθυνση γιατί ε, δίνει τη δυνατότητα σε αρχές ανταγωνισμού να αντιμετωπίσουν τις παραβάσεις. Όμως έχει ένα, ένα μειονέκτημα σημαντικό η πρόταση, δηλαδή ε, κάτι που απειλεί ολόκληρη την ε, θεσμική αρχιτεκτονική ε, του νέου καθεστώτες και την ευημερία του καταναλωτή. Ο βασικός στόχος του ευρωπαϊκού δικαίου ανταγωνισμού, οι συλλογικές αποζημιώσεις γίνονται μόνο σε μη υποχρεωτική βάση. Τα δικαιώματα του ανταγωνισμού ε, δεν εξασφαλίζονται εξίσου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το να υπάρχει ε, ένας ε, μηχανισμός σε περίπτωση σε περίπτωση ζημιών σε περιπτώσεις αντιτράστ μπορεί να έχει μερικές φορές κάτι, κάποιο ε, αποτέλεσμα κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα αδικαιολόγητο για κάποιου άλλους. Κάτι που σημαίνει μικρότερη προστασία για τους καταναλωτές. Αυτό σημαίνει forum shopping αθέμητο και αθέμητο αθέμητες αγορές. Αν θέλουμε να υπάρχει μία ισότιμη ε, μεταχείριση για όλους... Στην ενιαία αγορά θα πρέπει να εναρμονίσουμε τέτοια ζητήματα συλλογικών παρεμβάσεων. Γι' αυτό λοιπόν Χαιρόμαστε ιδιαίτερως που το σχέδιο γνωμοδότησης ε, θέτει λοιπόν το θέμα αυτό και επιπλέον ε, προβλέπει τέτοιους μηχανισμούς ε, και μείωση του κόστους βέβαια για τέτοιους αδύναμους ενάγοντες σύμφωνα με, τα, με τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής μας. Τέλος, όντως, είναι πολύ περίπλοκο το αντικείμενο της οδηγίας αυτή σε ό,τι αφορά τα μέτρα αντιτράστ και αυτό περιλαμβάνει την διάδραση μεταξύ της ιδιωτικής και δημόσιας επιβολής του δικαίου. Η δημόσια λοιπόν επιβολή του δικαίου χρειάζεται και την ιδιωτική ε, επιβολή του δικαίου προκειμένου να δρά ως αντικίνητρο και προφανώς χρειάζεται μια δυναμική δημόσια εφαρμογή γιατί υπάρχει η διάδραση σε ό,τι αφορά με τα θέματα αυτά που δεν ε, μπορεί να συνεπάρξει με τέτοια προγράμματα. Γι' αυτό λοιπόν τα προγράμματα αυτά ε, είναι σημαντικά σε ό,τι αφορά τα θύματα κατά, σε πρώτη, από πρώτη άποψη και γι' αυτό λοιπόν ε, οι τροπολογίες της κυρίας Ράπτη ε, προσπαθούν ακριβώς αυτό να πετύχουν, την καλύτερη ισορροπία μεταξύ των εγγυήσεων και των ενδιαφερόντων και συμφερόντων των καταναλωτών της ενίας αγοράς και της κοινωνίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας... Ευχαριστώ συνάδελφε. Το λόγο τον έχει ζητήσει από πλευράς πρασίνων ο εκπρόσωπος. Σας ευχαριστώ, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Θα χαιρόμουν ιδιαίτερος αν καταφέρναμε να βρούμε μια συμβαστική λύση και να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Γιατί νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τι ε, συλλογικέ αυτές αγωγέ, δεν έχει κανένα νόημα να είναι κανεί αμετακίνητο. Άρα λοιπόν όντω χρειάζεται συμβιβασμό. Να δούμε πως κάποιος άλλος θα επιθυμεί το λόγο. Όχι. Ο κύριος Γιούμπιτ από την Επιτροπή έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα τους βουλευτές που πήραν το λόγο. Σημείωσα διάφορα σημεία τα οποία ετήχθησαν. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τις συλλογικέ αγωγές. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηρτήσε μία πολιτική και την παρουσίασε ως εναλλακτική λύση για να, για να διευθετεί το θέμα αυτό με οριζόντια. Αυτή ήταν και η άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως γνωρίζετε. Οι εμπλεκόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μας είπαν ότι το θέμα αυτό είναι οριζόντιο και αυτό είναι σημαντικό σε ό,τι αφορά θέματα ανταγωνισμού. Και γι' αυτό λοιπόν θα έπρεπε να αποφευθεί ο κατακαιρματισμός μέσω των εθνικών μέτρων. Και θα ξέρετε ότι πολλά κρατημέλη συζητούν το φόρουμ ε, συλλογικών συμβάσεων, συλλογικών αγωγών που θέλουν να εισαγάγουν και το Ηνωμένο Βασίλειο και το Βέλγιο. Άρα μας είπαν ότι ας περιμένουμε μέχρι ότου αποδειχτεί περίτρανα και ανδιαφυσβήτητα ότι το ευρωπαϊκό επίπεδο είναι το καλύτερο επίπεδο αντιμετώπιση των συστημάτων αυτών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε να προστατεύσουμε με τον καλύτερο τρόπο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και θεωρούμε ότι με την οδηγία θα βελτιωθεί σημαντικά η δυνατότητα αποζημίωσης των πιο αδύναμων αυτών μερών. Αναφέρθηκαν και οι διαδικασίες επιβολής κυρώσεων. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι τι γίνεται με τις έμεσες αγορές, το οποίο αναφέρθηκε και από τον κύριο Σμιτ και από άλλους. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να έχουν πραγματικές δυνατότητες. Να δούμε για παράδειγμα το παράδειγμα διαφόρων καρτέλ σε ό,τι αφορά παραγωγούς ε, βιταμινών, ζωοτροφών, προϊόντων κρέατος αν λοιπόν διαπιστωθεί όντω παραβίαση και υπερβολική τιμολόγηση ω απορία αυτή, θεωρούμε ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε με την πρότασή μα μια πρόβλεψη σε ό,τι αφορά την υπερτιμολόγηση και το να αναστραφεί το βάρος αποδεξής. Γιατί προφανώς η ενάγοντες δεν μπορούν να ξέρουν τι ακριβώς έγινε και πώς προέκυψε αυτή η υπερτιμολόγηση σε μια λυσίδα την οποία δεν γνωρίζουν. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό το κομμάτι. Ένα άλλο θέμα το οποίο συζητήθηκε είναι η ισορροπία μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής εφαρμογής. Φυσικά, απότερο σκοπό είναι να υπάρχουν και τα δύο σκέλη δυναμικά. Βελτιώνοντας την ε, κατάσταση λοιπόν για τους ανάγοντες, δεν θέλουμε να θέσουμε να αμφιβόλο την δημόσια εφαρμογή. Και σε ό,τι αφορά α, όσους αντιμετωπίζονται με επίκη τρόπο. Υπάρχουν ορισμένα όρια μέσα στα οποία μπορούμε να δράσουμε και πιστεύουμε ότι η πρότασή μας η δημιουργία δηλαδή ενός μαύρου καταλόγου μιας μαύρη λίστας είναι ο σωστό τρόπος να αντιμετωπίσουμε το θέμα που δίνει η νομική σαφήνεια και σε όσου ζητούν επίοικια και στα άλλα μέρη για το τι είναι προσβάσιμο και το τι δεν είναι προσβάσιμο και υπό ποιου όρου. Νομίζω ότι στο σημείο αυτό θα σταματήσω. Ευχαριστούμε. Ο εισηγητής κύριος Μήθα έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τα σχόλια που κάνετε ασφαλώς. Ασφαλώς ε, ξέρω πόσο ευαίσθητο είναι το θέμα αυτό. Το γνωρίζω. Και γνωρίζω ότι έχουμε και διαφορετική αντιμετώπιση και σε τελική ανάλυση ασφαλώς θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση. Αυτό το αντιλαμβάνομαι. Καταλαβαίνω βεβαίω και τα επιχειρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ όμως πάντα θεωρούσα ότι το θέμα αυτό, ότι το σώμα μας είναι πολιτικό στη φύση του. Εγώ είμαι πολιτικός. Άρα η άποψή μου και αυτά που μπορεί να κάνει η Επιτροπή δεν είναι μόνο να νομοθετεί, να παρουσιάζει τα γεγονότα, αλλά και το να παράσχει ένα όραμα. Και εγώ νομίζω ότι σε αυτό εστερούμε για το τι θέλουμε, για το τι μέτρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και γι' αυτό, γι' αυτό προσέθεσα κάποιες επιπλέον προτάσεις, όχι για να σας ε, ενοχλήσω, Άντρια ε, ε, Ίσως λιγάκι, αλλά όχι πολύ. Και όχι σας προσωπικά. Εγώ συζήτησα εκτενώς με τους Γερμανούς συναδέλφους στην ομάδα μου και πραγματικά δεν καταλαβαίνω τα επιχειρήματα που προβάλλουν. Ασφαλώς και είναι μεγάλη χώρα Γερμανία, Ασφαλώς και μπορούμε να υιοθετήσουμε τους δικούς σας κανόνες. Δεν νομίζω όμως ότι με τον τρόπο αυτό οδηγούμε στην Ευρώπη. Αν θέλουμε, και ελπίζω, ελπίζω να με υποστηρίξει εδώ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν θέλουμε πραγματικά να υπάρχει μια ενιαία αγορά φιλική προς τον καταναλωτή, μα χρειαζόμαστε κάποιον μηχανισμό, κάποια μέσα τέτοια. Εγώ νομίζω ότι από το 99 που ήρθα στο κοινοβούλιο εδώ τα συζητάμε αυτά. Και υπάρχουν πολλά επιχειρήματα ότι α, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα, χρειάζεται χρόνο, του χρόνου ίσως. Αυτή είναι η βασική μου λοιπόν τοποθέτηση για τα υπόλοιπα θέματα. Είναι λεπτομέρειες, ξέρετε. Αλλά όπως ξέρετε και ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Και θεωρώ λοιπόν ότι χρειάζεται μια ισορροπία. Κατανοώ τα επιχειρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε κάποιους ωστόσο τομείς θεωρώ ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βάλουμε τον καταναλωτή και τα συμφέροντα του καταναλωτή πάνω από όλα. Και μπορούμε να διαφωνούμε ασφαλώς και να λέμε ότι «Α, κοιτάξτε, αυτό δεν είναι προς το συμφέρον του καταναλωτή». Ενδεχομένως, αυτό ναι. Αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να είναι πλήρης και εντελεχής η συζήτηση σε σχέση με το τι είναι το καλύτερο, ποια είναι τα καλύτερα μέτρα για τον καταναλωτή προκειμένου να δράσει, να αντιδράσει και άρα θεωρώ ότι χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση σε ό,τι αφορά όλες αυτές τις διαφορετικές προτάσεις και φυσικά σε τελική ανάλυση σύμφωνο Ασφαλώς και θα βρούμε κάποιο συμβασμό. Βεβαίως. Εγώ θα υπερψηφίσω τη δική μου τοποθέτηση Ελπίζω και εσείς αυτό να κάνετε. Ελπίζω και ο κύριος Σβάμπ να υπερψηφίσει και θα υπερψηφίσω ασφαλώς και την έκθεση του κυρίου Σβάμπ στην Επιτροπή ΕΚΟΝ. Έτσι είπαν τα πράγματα εδώ. Και Νομίζω ότι το θέμα των συλλογικών αγωγών μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Εγώ είμαι φιλελεύθερος, δεν θέλω να υπάρχει τόσο μεγάλος λογικό χαρακτήρας στα πάντα, αλλά νομίζω ότι σε κάποιες περιπτώσεις είναι κανείς πολύ μόνος και μπορεί να βοηθηθεί από τίποτε. Άρα χρειάζονται σε κάποιες περιπτώσεις συλλογικά μέτρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, λέει ο Πρόεδρος. Ποιο άλλο. Α, μισό λεπτό. Να σας ενημερώσω για κάτι. 18 Οκτωβρίου τελευταία προθεσμία για τις τροπολογίες. Αυτό θα ήθελα να σας πω. Στη συνέχεια το σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. Εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υποπίεση στην αγορά. Ε, έχει λάβει το λόγο και έχει φραστεί ο συνάδελφος Ιωάμπαμ και γι' αυτό το λόγο θα μπορούσε να λάβει ο σκιώδης εισηγητής και αν ο συνάδελφος Ζουάμπ όμως θα ήθελε, θα επιθυμούσε το λόγο, εντάξει. Έχει τη δυνατότητα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αλλά μίλησα, μίλησα στην εισαγωγή μου. Δεν θέλω λοιπόν να προσθέσω ιδιαίτερα πράγματα, ούτε να χάσουμε χρόνο με το θέμα αυτό. Τα θέματα που έθεσα τα επιπλέον ισχύουν όπως ισχύαν και για το σημείο 3 της σημερινής διάταξης. Άρα θα ήθελα, αν θέλετε, να μην ε, χρειαστεί να δώσετε το λόγο στην κυρία Ροϊτοβά, η οποία είναι η συγκεκριά μα, γιατί ουσιαστικά εγώ την εκπρόσωπο δεν είναι εδώ και θα χρειαστεί να επαναλάβω ακριβώ τα ίδια που είπα και προηγουμένω. Also ich kann es auch wieder mal ganz kurz machen. Θα είμαι και πάλι πάρα πολύ σύντομη. Υποστηρίζουμε τις προτάσεις, το ανακοινώσαμε στην κυρία Ρόιτοβα, προέρχονται από το Liment Packet, στο οποίο ήμουν και η συγγήτρια και αυτό λοιπόν το θέμα φαίνεται ότι επιτέλους, επιτέλους προχωράει. Για να κλείσουμε τη συζήτηση για το Lyman Package. Ελπίζω και η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων να τοποθετηθεί, να υποβάλει την γνωματοτησή τη, προκειμένου το συντομότερο δυνατόν να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό. Ο κύριος Φόξ έχει το λόγο. Πρόεδρε, πολύ μας χαροποιεί που προχωράει αυτό το θέμα και δεν χρειάζεται οποιοδήποτε άλλο σχόλιο. took everyone by surprise, didn't it? Κυρία Ζήρο, από την Επιτροπή έχει το λόγο τώρα. Ο κύριος, ευχαριστώ, ο Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να κάνουμε κάποια σχόλια για την έκθεση. Θα θέλαμε σε πρώτη φάση να σας ευχαριστήσουμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Ρόιτοβα για την έκθεση. Στην ε, πράξη, να, ε, ουσιαστικά συμφωνούμε με τα στοιχεία, όλα τα στοιχεία. Κάποια, ωστόσο, θεωρούμε ότι δεν είναι τόσο ουσιώδη, κάποια είναι ίσως ε, υπερβολικά ως διατυπώσεις, μίλω στην 23, 30, 39, 43 και 44 τροπολογίες αυτές. Στην 23 προτείνεται να εισαχθεί μια πρόταση που θα μιλάει upon a duly justified request of the content authorities με την δέουσα αίτηση των σχετικών αρχών. 23.6 για το άρθρο 6. Μιλάμε για τις υποχρεώσεις του ε, κατασκευαστή. Με το κείμενο λοιπόν που προτείνουμε είναι το ίδιο του πακέτου. Εδώ πέρα τη ζητάμε να έχουν ενεργό ρόλο η, καταγωγή, η παραγωγή σε ό,τι αφορά τις ε, επιθεωρήσεις και όχι μόνο όταν του ζητείτε αυτό από τις αρμόδιες αρχές. Στην 30 ε, τώρα. 14 άρθρο, παράγραφος 4. Μιλάμε για το γλωσσικό καθεστώς. Φυσικά συμφωνούμε πάντα ότι το γλωσσικό καθεστώς ε, πρέπει να περιλαμβάνει γλώσσες που να καταλαβαίνουν οι καταναλωτές. Ωστόσο, εδώ σε αυτό το άρθρο μιλάμε για τη σχέση μεταξύ των ε, υπηρεσιών αξιολόγησης ε, συμμόρφωσης και των καταναλωτών και των παρασκευαστών και των ε, καταναλωτών. Οι καταναλωτές όμως δεν επεμβαίνουν σε αυτό το θέμα. Τα έγγραφα τα οποία υποβάλλουν δεν προορίζονται για τους καταναλωτές, μόνο για τους κατασκευαστές και για τις σχετικές αρχές των κρατών μελών. Για την τροπολογία 32, και αυτό σχετίζεται και με την τροπολογία 43 και 44, προτείνεται στο άρθρο 26 αντί να αναφέρεται το presumption of conformity να αναφέρεται presumption of conformity of the notified bodies. Και επειδή υπάρχουν ιδιαιτερότητε στην νομοθεσία, δεν είναι μόνο τα οι κοινοποίηση που κάνουν αξιολόγηση. Υπάρχουν τρει ομάδε ομάδες. Οι υπηρεσίε κοινοποίηση, οι αναγνωρισμένε οργανώσει τρίτων μερών και μία ομάδα που ονομάζεται επιθεωρητέ χρηστών. Άρα δεν μπορούμε να αναφερόμαστε μόνο σε αυτά τα notified bodies. Ίσως θα μπορούσαμε να αναφέρουμε κάτι πιο γενικό. Conformity Assessment Bodies, 43 και 44 τώρα τροπολογίες και πάλι γίνεται τέτοια αναφορά στα Notified Bodies, να αναφέρουμε στα Conformity Assessment Bodies υπηρεσίες ελέγχου συμμόρφωση. Θεωρούμε λοιπόν ότι δεν είναι θέματα ουσίας αυτά, είναι θέματα επί των οποίων πολύ γρήγορα μπορούμε να αποφασίσουμε και κατά τα άλλα δεν έχουμε οποιοδήποτε άλλο σημαντικό πρόβλημα. Νομίζουμε λοιπόν ότι θα καταφέρουμε να συμφωνήσουμε χωρίς κανένα πρόβλημα από το κειμένο. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Ήδη έχουν εκφράσει την άποψή τους οι συντονιστές και συμφώνησαν για την απλοποιημένη διαδικασία. Η εισηγήτρια και μόνο θα μπορούσε να υποβάλει τροπολογίες. Άρα λοιπόν προχωράμε και στις 25 Νοεμβρίου για την ψηφοφορία. Το σημείο 7 τώρα. Είναι η έκθεση που αφορά την ασφάλεια καταναλωτικών προϊόντων. Η κυρία Σαλδεμός είναι η εισηγήτρια. Να περιμένουμε πέντε λεπτά για να έρθει η συνάδελφος. Συμφωνείτε έτσι, βέβαια.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 Μπορούμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας, έτσι. Ήλθε εδώ η συνάδελφος. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Άργησα λίγο, συγγνώμη σας παρουσιάζω τις ε, συμβαστικές τροπολογίες εντάχει και θα σας ενημερώσω για το που βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά το CPSA. Να ευχαριστήσω τους κοιόδους εισηγητές καταρχής για τις καλές συναντήσεις που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Νομίζω ότι οι διαπραγματεύσεις προχωρούν με καλό τρόπο. Πιστεύω δε ότι θα είμαστε σε θέση να πετύχουμε καλούς εμβιβασμούς συμβάλλοντας ε, καλά σε αυτή την νομοθεσία για την ασφάλεια των προϊόντων. Εννέα διαφορετικούς συμβαστικούς ε, Συμβαστικέ προτάσει έχω κάνει. Δεν θα τι ε, εξετάσω ενδελεχώ. Θα σα παρουσιάσω μόνο τα θέματα. Καταρχά, νομίζω καταφέραμε να βρούμε συμβιβασμό για τον ορισμό της χρήσης των προϊόντων σε σχέση με τις υπηρεσίες για επίσης συμβασμό για τα προϊόντα που απευθύνονται στα παιδιά. Δεν έχουμε ολοκληρώσει απόλυτα την πρόταση αυτή, αλλά κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Όλοι συμφωνούν ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις τώρα. Συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν να υπάρχει ίδια διατύπωση και στις ε, δύο νομοθεσίες, και στο CPSA και στο NSA. Νομίζω λοιπόν ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να υπάρξει η διατύπωση και σε ό,τι αφορά τις κυρώσει. Εδώ λοιπόν πιστεύουμε όλοι ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ισχυρή, στεναρή διατύπωση για να ξεκαθαρίζεται ότι υπάρχει ευθύνη του, κα, του παρασκευαστή, του κατασκευαστή και αν δεν τηρείται θα πρέπει να υπάρχει κάποιο κόστος ως απορία. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες όμως στην παρούσα φάση. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλές ε, οι συζητήσεις για το CE+, το CE συν. Δεν έχουμε καταλήξει σε κάποια λύση. Σημειώνω ωστόσο ότι οι συνάδελφοι συμφωνούν ότι το σήμα CE όπως χρησιμοποιείται σήμερα δεν ε, λειτουργεί σωστά. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό αποτελεί ένα καλό σημείο κίνηση για να βρούμε μια μελλοντική λύση. Δεν έχουμε βρει ακόμα τη λύση αυτή σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη διατύπωση αλλά θεωρώ και ελπίζω ότι ως εθελούσιο σύστημα είναι χρήσιμο για τους καταναλωτές και για τις καλές επιχειρήσεις, τις καλές εταιρείες ε, της εσωτερικής αγοράς. Συμφωνία επίσης έχουμε για την αρχή της πρόληψης σε ό,τι αφορά τη συμπερίληψη της αρχής αυτής της νομοθεσίας. Α, προσπαθούμε να βρούμε το πιο κατάλληλο σημείο για να συμπεριληφθεί τώρα το σημείο αυτό Έγιναν συζητήσεις επίσης ε, για τον κανονισμό για το δικτύο ασφαλείας. Συμφωνούμε όλοι ότι το πιο σημαντικό στοιχείο είναι να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχουν παραθυράκια. Δεν θέλουμε όμως να κινηθούμε πέρα από αυτά. Ψάχνουμε να βρούμε μια καλή διατύπωση για να κλείσουμε τα κενά. Προσπαθούμε να βρούμε συμβιβασμούς επίσης για τις ε, λογικές ε, λογικούς όρους, προβλέψιμους όρους για τον ευάλωτο καταναλωτή. Νομίζω ότι θα καταφέρουμε να βρούμε μια λύση. Καλό θα είναι να μην επισέλθουμε σε υπερβολικέ λεπτομέρειε. Το μεγαλύτερο θέμα το οποίο συζητήσαμε την προηγούμενη φορά ήταν η υποχρέωση του οικονομικού operator. Ως τώρα υπάρχει συμφωνία ότι θα πρέπει να βρεθεί μια διατύπωση που θα ακολουθεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό είναι καλό γιατί στην περίπτωση αυτή δεν αποδυναμώνουμε τις υποχρεώσεις για τους οικονομικούς διαχειριστές. Αλλά θα μπορέσουμε να είμαστε πιο ακριβείς σε ό,τι αφορά κάποιες υποχρεώσεις για να μην υπάρχει παρανόηση. Να είναι σαφές τι είδους υποχρεώσεις έχει ο κάθε διαχειριστής σε κάθε τμήμα της αλυσίδας. Και εδώ λοιπόν θεωρώ ότι θα βρούμε μια λύση. Αυτές είναι λοιπόν κάποιες από τις τροπολογίες. Τέλος σε ζητούμε τι είδου εξαιρέσει από τι ε, υποχρεώσει του οικονομικού operator θα πρέπει να προβλέπονται. Ω τώρα λοιπόν δεν έχει ολοκληρωθεί το στάδιο αυτό. Νομίζω όμω ότι κινείται προ τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ και πάλι του κοιόδε εισηγητέ. Ε, δύο θέματα ακόμα ήθελα να αναφέρω. Ένα είναι ότι πέρα από του συμβιβασμού αυτού είναι σημαντικό, θεωρώ, να υπάρχει και στο CPSR και στο MSR για μια ενδιάμεση βάση δεδομένων για τις σοσιαλιστές και δημοκράτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει το εργαλείο αυτό. Είναι λοιπόν μια κόκκινη γραμμή. Με κάποιο τρόπο να συμπεριληφθεί αυτό. Τελευταίο στοιχείο που θα ήθελα να αναφέρω προς τους συναδέλφου. είναι το εξή. Δεν προσπαθούμε να συμβιβαστούμε για τη διατύπωση, για το άρθρο 7, για το σήμα Made in παρασκευάζεται σε ποια χώρα. Κατά πάσα πιθανότητα λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει ξεχωριστή ψηφοφορία στην Επιτροπή μας εδώ, στην Επιτροπή Προστασίας του καταναλωτή, γιατί διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε κάποια βάση επί της οποίας θα μπορούσαμε να βρούμε συμβιβασμό. Υπήρχαν δύο αντίθετες απόψεις, άρα η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ξεχωριστή ψηφοφορία. Αλλά τα υπόλοιπα κινούνται προς το εμπρός και είμαι αισιόδοξη ότι θα υπάρχει καλό, θα σημειώσουμε καλό αποτέλεσμα στην ψηφοφορία στα τέλη της εβδομάδας. Σας ευχαριστώ. Ο, ο πρόεδρος Ευχαριστώ πρόεδρε, δεν μιλάω εξ μου, μιλάω εξ ονόματος της κυρίας είναι η οποία δυστυχώς τέτοια ώρα σήμερα δεν μπόρεσε να παρευρεθεί και αν μου επιτρέψουν οι συνάδελφοι να πω και δύο λόγια εξ ονόματος δικού μου. Καταρχάς λοιπόν, εξ ονόματος της εισηγήτριάς μας, η οποία ασφαλώς καταρχάς ευχαριστεί όλους τους συναδέλφους που συνέδραμαν στην εξέβρεση συμβιβαστικών ε, λύσεων στην παρούσα οδηγία. Σας ευχαριστεί λοιπόν γιατί θεωρεί πολλά είναι πάρα πολύ επικοδομητικά, πολύ ωφέλιμα και ε, βελτιώνουν το αποτέλεσμα. Στους κοιόδες εισηγητές και στην Επιτροπή έχει υποβάλει 12 συμβιβαστικέ τροπολογίες που καλύπτουν όλα τα τμήματα της πρότασης και ενδεχομένως να προσθεθούν και άλλες συμβαστικές προτάσεις σήμερα το βράδυ, γιατί σήμερα το μεσημέρι γίνεται τεχνική συνάντηση των σχετικών υπαλλήλων. Η συναδελφός λοιπόν Πιετικάινεν μου ζήτησε να σας παρουσιάσω κάποιες ε, τροπολογίες. για να υπάρχει η βεβαιότητα ότι όλοι όσοι συμμετείχαν ξέρουν τι εννοείται. Γι' αυτό λοιπόν θα σας τα παρουσιάσω αυτά στα αγγλικά. Καταρχάς το θέμα είναι η διάκριση μεταξύ online και offline. Ο πρώτος η τροπολογία συμβαστική έχει σκοπό να καλύπτει η νομοθεσία όλα τα θέματα, ανεξάρτητα από το κανάλι διανομής. Ε, Ζητείτε λοιπόν διευκρίνηση προκειμένου ο κανονισμός να ισχύει και online και offline και θα πρέπει να υπάρχει ψηφιακός αλλά και φυσικός έλεγχος. Η διατύπωση του MLF προέρχεται μάλλον από το MLF σε ό,τι αφορά τα άρθρα για τα πυροτεχνικά ζητήματα. Ζητείται λοιπόν καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να διευκρινιστεί ο ρόλος της, ε, του ηλεκτρικού, ηλεκτρονικού εμπορίου μπορεί να είναι αντίθετο με το επιθυμητό αποτέλεσμα αν θέλαμε να προσθέσουμε online και offline σε μία τυχαία επιλογή άρθρων και αιτηλογικών σχέσεων. Γιατί έτσι θα σκεφτόταν κανεί ότι μπορεί να μην ισχύει κάτι παρόμοιο όπου δεν υπήρχε η διπλή αυτή αναφορά. Και δεν θα ήταν σαφέ τι θα γίνει με τι μελλοντικέ αλυσίδε διανομή. Δεύτερο σημαντικό θέμα, οι κυρώσει. Το Κοινοβουλίο ζήτησε κάτι που θα δράσει αποτρεπτικά ήδη στο ψήφισμα του 2011. Θα πρέπει λοιπόν να είναι ε, βαριά τα οικονομικά αντικίνητρα και κυρώσεις για αυτούς οι οποίοι θελημένα εισαγάγουν επικίνδυνα ή μη συμμορφούμενα προϊόντα στην ενιαία αγορά. Επίσης, να εισαχθούν πιο ε, δυναμικές διατάξεις σε ό,τι αφορά τα, τις κυρώσεις σε σχέση με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πρόταση επιτάπητος ε, έχει να κάνει με τέτοια θέματα κυρώσεων. Ωστόσο, ε, αντί να συνδεθεί το θέμα των κυρώσεων με τον προηγούμενο κύκλο ε, εργασιών, ίσως ήταν πιο σωστό να συνδεθεί με τις πωλήσει του εκάστοτε προϊόντος, γιατί μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να πρόκειται για μικρούς ή καινούριους ε, ε, πολιτές κατασκευαστές οι οποίοι δεν έχουν ε, παλαιό κύκλο εργασιών και έτσι θα μπορούσαμε να επιβάλλουμε κυρώσεις βάσει του κύκλου εργασιών. Ένα τρίτο θέμα είναι η σχέση μεταξύ μη συμμόρφωσης και κινδύνου. Έχουμε δύο ξεχωριστούς ορισμούς του μη συμμορφούμενου προϊόντος και του προϊόντος που παρουσιάζει κίνδυνο. Προτείνεται ότι η διάκριση αυτή σε ό,τι αφορά τον ορισμό του μη συμμορφούμενου προϊόντος να συμπεριλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις μη συμμορφούμενων προϊόντων. Δηλαδή και εναρμονισμένων και μη εναρμονισμένων προϊόντων. Το θέμα του ορισμού συνδέεται με το ρόλο της RAPEX αφενός και του ICMSMS αφετέρου. Η εισηγήτρια ασφαλώς παραμένει ανοιχτή για τα σχόλιά σας και όπως σας είπα πρόεδρε, όπως θα παρουσιάσω και κάποια σημεία, όχι εξ ονόματος της κυρίας Πιατικάνεν πλέον, αλλά να μιλήσω εξ ονόματός μου. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν υπάρχει πρόταση συμβαστική για το άρθρο 7 σε ό,τι αφορά την πρόταση του, για το made in. Τρεις φορές ήδη στο Συμβούλιο, να το θυμόμαστε, έχει απορριφθεί αυτή η πρόταση, όλος χειρός. Δεν βλέπω λοιπόν γιατί θα διέφερε η κατάσταση σε μια τέταρτη πρόταση. Εγώ προσωπικά λοιπόν είμαι της άποψης ότι μη συμβιβαστική πρόταση θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξέβρεση συμβιβασμού με το Συμβούλιο παρά να παραμείνει η πρόταση όσο έχει στο άρθρο 7. Δεύτερη παρατήρηση για αυτά που είπε η κυρία Σαλτεμόζα για το σήμα C+, συν. Έχουμε δει πρόσφατα παρουσιαστήκε το σκάνδαλο με τα επιτεύγματα για εγχειρήσεις ε, στήθους και πρέπει να πω ότι γενικά είμαι πάρα πολύ επικριτικό σε ό,τι αφορά αυτή την ιδέα. Αν είμαστε όμως έτοιμοι να αποδεχτούμε το σύστημα αυτό, να γίνει επιπρόσθετα με τη χρήση του σήματος CE, το CE+, μετά από κάποιον έλεγχο. Αλλά θεωρώ ότι αυτό που έχουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή ε, δεν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι αποδεδειγμένο αυτό. Η αρχή της πρόληψης ε, νομίζω ότι επιλύεται στο πεδίο εφαρμογής, πολύ αποτελεσματικό. Ευχαριστώ την κυρία Σολτεμόζα και η συμπερίληψη των ε, συγκεκριμένων αναγκών των ευάλωτων καταναλωτών τα πράγματα δεν είναι ιδανικά, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρό το αποτέλεσμα και καλό το αποτέλεσμα και σας ευχαριστώ λοιπόν. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε. Για να δούμε τώρα αν υπάρχει κάποιος άλλος που θα επιθυμούσε το λόγο. Τι ζήτησε ο κύριος Φόξ, ζήτησε τον λόγο η κυρία πριν από τις ε, υπόλοιπους γιατί θα πρέπει επιγόντως να αναχωρήσει. Α, λοιπόν η κυρία Φόξ θα λάβει το λόγο και μετά οι υπόλοιποι. Α, ο κύριος, συγγνώμη, ο κύριος, ο κύριος. Στις ώρα στις ταγματικές υποθέσεις ε, ψηφίζουμε για την ε, μοναδική έδρα ε, οπότε προσπαθώ να ψηφίσουμε όλες τις γνωμοδοτήσεις ε, που θα ε, εξοικονομήσουν πολλά λεφτά φορολογουμένων, άμα έχουμε μία μόνο έδρα. Τέλος πάντων, σε σχέση με την εποπτεία της αγοράς και το σχετικό κανονισμό, τα σχόλιά μου έχουν να κάνουν μόνο με τις κυρώσεις και έχει να κάνει, έχουν να κάνουν και με αυτό που είπε η κυρία Σαλντεμόσε. Νομίζω ότι οι προτάσεις μας εδώ είναι αυθαίρετες και εντελώς δεν υπάρχουν στοιχεία δηλαδή. Θα έπρεπε οι κυρώσει να είναι αποτρεπτικέ ε, και αναλογικέ. Αν το υπερβούμε να μπερδεύουμε τα πράγματα και να λέμε ότι σε αυτή την περίπτωση πρέπει να χάνει με τα κέρδη, αλλά σε μια άλλη περίπτωση, αν δεν ε, υπάρχει συμμόρφωση, αν δεν υπάρχει κίνδυνο, θα έπρεπε να υπάρχει το τάδε επίπεδο κυρώσεων. Προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν οι συνάδελφοι, αλλά τελικά θα είναι επιπόλαιη η νομοθέτηση. Α μείνουμε με αυτήν την καλά, πολύ δοκιμασμένη ε, φόρμουλα, δηλαδή να είναι αποτρεπτικέ οι κυρώσεις και να αφήσουμε στα κράτη-μέλη τα υπόλοιπα, γιατί διαφορετικά δημιουργούμε ένα νομοθετικό χάος. Τώρα, σε σχέση με τα σχόλια της κυρίας Σαλντεμόσε, ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια της. Ε, εξακολουθώ να ανησυχώ με, το, με την ε, με την αγορά, με, το, με τη σήμανση του, την κοινοτική. Τα εμφυτεύματα αυτά είχαν, όλοι αυτό το, είχαν όλο αυτό το σήμα. Αν κάποιος είχε κάνει παραποίηση, δηλαδή θα είχε καμία διαφορά αυτό, το αν είχε κοινοτικό σήμα ή όχι. Όχι, δεν θα είχε τελικά για τον άνθρωπο που θα είχε το εμφύτευμα. Λοιπόν, ας μην γελιόμαστε. Εμείς μπορεί να νιώθουμε καλύτερα ότι κάτι κάναμε με αυτά που λέμε, αλλά δεν προστατεύουμε όντω του καταναλωτές. Δημιουργούμε ακόμη ένα εμπόδιο, το οποίο πρέπει να το υπερβούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μερικές ακόμη ανησυχίε έχω. Η νομοθέτηση για ε, τις της ε, δικαστικό διορισμό ε, των υπευθύνων εποπτείας αγοράς. Δεν νομίζω ότι είναι δική δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό. Υπάρχουν ε, άκαμπτοι κανόνες που δημιουργούν επιπλέον γραφειοκρατία αν ε, κατασκευάζει κανείς ένα αυτοκίνητο, ελπίζω να κρατάει τη σχετική τεκμηρίωση για πάνω από 10 χρόνια. Αν όμως κάνει όμως ένα κύβο ζάχαρης ή ένα ποτήρι ή ένα μολύβι, νομίζω ότι το να έχουμε τόσο πολύ καιρό να κρατάμε τα έγγραφα δεν χρειάζεται. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να νομοθετούμε καλύτερα όμως, όταν βλέπω τις συμβιβαστικές τροπολογίες, βλέπω επαναλαμβανόμενη άχρηστη διατύπωση που απλό σκοπό έχει να χαροποιήσει όλο τον κόσμο. Και τελικά θα φτιάσουμε σε ένα κείμενο το οποίο είναι υπερβολικά λεπτομερές, δυσανάγνωστο και πολύ δύσκολο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν νομικό τμήμα να το κατανοήσουν. Έχω χρησιμοποιήσει αυτή την αναλογία στο παρελθόν. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο και όλοι βάλουμε, βάζουμε το δικό μας στολίδι πάνω για να είμαστε ευχαριστημένοι και το αποτέλεσμα ήταν, είναι μια ιδέα που δεν έχει κανένα απολύτως, ε, καμιά απολύτως συνέχεια. Δηλαδή, ε, το να λέμε τι θέλουμε να κάνουμε είναι απλώ μια θήλωση προθέσεων. Εδώ όμω νομοθετούμε. Δεν τα λέμε απλά, τα νομοθετούμε κιόλα. Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Γιατί νομίζω ότι το να βάζουμε τόσου πολλού συμβιβασμού, όλο και περισσότερο προσθέτουμε, δυσκολεύοντα έτσι τη ζωή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Προσπαθούμε να βγούμε από μια κρίση, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε θέσει εργασία και αυτή η νομοθεσία θα έπρεπε να διευκολύνει τα πράγματα, να απλοποιεί όταν διαβάζει κανείς τις συμβιβαστικές τροπολογίες είναι τρομερά περίπλογες. Πώς είναι δυνατόν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν την νομοθεσία αυτή. Οπότε ευχαριστώ πολύ και, τον, ε, και τους, ε, και τους, εισηγητές, και τους εισηγητές ε, και τον εισηγητή και όσους κατέθεσαν τροπολογίες. Συγγνώμη αν φύγω σε πέντε λεπτά για να προσπαθήσω να περισσώσω κάποια χρήματα των φορολογουμένων. Σας ευχαριστώ και εσάς. Και τώρα ο κύριος Μπαλτάσαρ. Ναι, πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε σχετικά με την έκθεση αυτή. Που μπορώ να πω ότι έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα είναι δύσκολο το έργο και να προστατεύσουμε τους καταναλωτές. Γιατί τα διάφορα που προέκυψαν αυτά τα χρόνια αποτελούν μια μαρτυρία ότι κυκλοφορούν στην Ευρώπη πολλά προϊόντα που δεν είναι σίγουρα και δεν γνωρίζουμε ούτε καν την προέλευσή τους. Άρα λοιπόν είναι βάσιμη αυτή η υποψήφια και καλό είναι υπάρχει μια οδηγία, ένας κανονισμός, κάτι πάντων που να το εξετάζει αυτό. Και επίσης να αποφύγουμε αυτή η ρύθμιση να αποτελεί γραφειοκρατικό εμπόδιο για τις εταιρείες. Πάντως καταβάλλεται προσπάθεια, εργαζόμαστε από κοινού και εύχομαι να πετύχουμε μία λύση θετική στο τέλος. Σχετικά με την συμβαστροπολογία 1, εκεί πετύχαμε μία λύση για την τροπολογία Fox καλό αυτό και ο συνάλφος θα μπορούσε να είναι κάπως περισσότερο αισιόδοξο. Για τη συμβαστική τροπολογία 2 τώρα, για τα ελκυστικά για τα παιδιά προϊόντα, τα μικρά μικρά παιδιά, εδώ θα πρέπει να βρούμε ένα ορισμό που να είναι περισσότερο ακριβής. Αλλά αυτή η ανάγκη να πετύχουμε ένα σαφή συγκεκριμένο ορισμό θα πρέπει να συνδυαστεί και με την ανάγκη να εξασφαλίζονται τα παιδάκια μας ε, στην αγορά προϊόντων, προϊόντων που απευθύνονται σε αυτά, τα παιδιά. Πάρα πάρα πολλά παραδείγματα παιχνιδιών υπάρχουν ε, από τοξικά προϊόντα, καθόλου σίγουρα χρωστικές ουσίες ε, με επικίνδυνα συστατικά αλλά λοιπόν χρειάζεται να βρούμε ένα ακριβέστερο ορισμό ταυτόχρονα με το να προστατεύσουμε την παιδιά για τις ε, ε ποινές, ας το πούμε έτσι. Το πετύχαμε να τα συνδυάσουμε αυτά και με την επαγρύπνηση στην αγορά και να δούμε στη συνέχεια. Εδώ υπάρχουν ε, διάφορες υποθέσεις για το δρόμο που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε για μια συμφωνία είναι να τονίσουμε καλύτερα τον προαιρετικό χαρακτήρα της α, μάρκας και να το θεωρήσουμε σαν ένα, κάποια ένδειξη της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων. Αν μια επιχείρηση αν το θεωρεί ότι τελικά αυτά που επιβάλλονται είναι υπερβολικά και ότι δεν τους επιστρέφεται το όφελος ε, στην πρόθεση της εταιρείας τους, έτσι κι αλλιώς είναι προαιρετικού χαρακτήρα, μη δεσμευτικού. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να πετύχουμε μια συμφωνία. Εντάξει, για την πρόληψη, καλό. Και για το δίκτυο ασφάλειας, η θέση μας είναι πλησιέστερη προς τη θέση της Επιτροπής. Και εδώ προσπαθούμε να πετύχουμε μία συμφωνία. Μία συμφωνία που να ικανοποιεί αυτό το κριτήριο, να μην αφήνει κένα, τμήματα που να μην καλύπτονται χωρίς όμως να δημιουργήσουμε και διαφορές όσον αφορά τη ρύθμιση και για την προστασία των ε, ευάλωτων καταναλωτών και εκεί που εργαζόμαστε για να πετύχουμε κάτι. Επίσης και το 8 Δέλτα 8 Β και επίσης τονίζουμε το ότι δεν θα πρέπει να επιβαρύνουμε τους διανομής ε, με πράγματα που δεν είναι αρμοδιότητές τους. Δηλαδή αν θα μπορούσε και να δοκιμάζει το προϊόν. Εντάξει το πολύ πολύ άντε να δει αν υπάρχουν οι βεβαιώσεις, οι εγγυήσει ε, που έχουμε καθορίσει για τους εισαγωγείς ε, και για τους ε, εμπόρους, αλλά όχι ήδη να δοκιμάζουν τα προϊόντα και ακόμα ορισμένες τεχνικής φύσεως πτυχές που θα πρέπει περισσότερο να διευκρινίσουμε για να πετύχουμε επαναλήψεις να λέμε πολλές φορές τα ίδια πράγματα και να δούμε το 8 με το 9 άρθρο, το ένα το άλλο, μήπως να τα συνδυάσουμε. Διαφορετικά κινδυνεύουμε να επαναλάβουμε αρκετές φορές την ίδια υποχρέωση. Για να δούμε τώρα με το πολυσυζητημένο θέμα του άρθρου 7. Οι θέσεις αυτές κάπως αποκλίνουν. και στο Συμβούλιο ιδιαίτερα έχει αλλάξει κατάσταση σε σχέση με προηγούμενες φορές. Είναι μια αντιπαράθεση κατά κάποιο τρόπο που δεν ε, χαρακτηρίζει την κατάσταση τους τυπικούς υπερασπιστές, ε, αλλά υπάρχει μια κάποια μεγαλύτερη βιστοποίηση για τα προϊόντα αυτά, και στις χώρες προέλευσης ε, και γι' αυτό ακριβώς ε, να που ισχύει μια αλληλεγγύη και μια σύγκληση που δεν περιμέναμε από την Γαλλία, την Πολωνία κλπ. Και που λένε ότι αυτό που έχει σημασία είναι η ανάγκη στην κυκλοφορία των προϊόντων ε, στην Ευρώπη να υπάρξει και η ένδειξη προέλευσης, χώρας προέλευσης. λοιπόν να το πούμε και αυτό καθαρά. Με τον Ανδρέα συμφωνώ ότι θα πρέπει να δούμε γιατί είναι περίπλοκο το θέμα και σίγουρα θα υπάρξει ένας τριμερής διάλογος για να πετύχουμε μια συμβιβαστική λύση. Επειδή όμως υπάρχει δυσκολία αυτές τις τελευταίες 48 ώρες πριν από την ψηφορία, δύσκολο να πετύχουμε μια συμφωνία. Να δούμε αν αυτόνομα με εκφραστεί το Κοινοβούλιο, τι γραμμή θα χαράξει και μετά θα δούμε πώς ε, θα προβληθεί αυτό στον τριμερή διάλογο με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Αλλά σε παρόμοιο θέμα θα πρέπει να έχουμε πιο συγκεκριμένη άποψη, σαφή και να ακουστεί έτσι και η γενική άποψη του Κοινοβουλίου μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Βαλτάσαρ, λέει ο πρόεδρος. Ποιος έχει το λόγο τώρα. Ε, αν μήπως επιθυμεί το λόγο. Ε, ναι. Νομίζω ότι υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που θα θέλουν να πούν κάτι και ίσως καλύτερα να συνοψίσω στο τέλος. Ε, Άρα λοιπόν από τους φιλελεύθερους ο Μάντελς να λάβει το λόγο, μια και εσείς δεν τον επιθυμείτε προς το παρόν. Ευχαριστώ. Κρίστελ, πάρα πολύ καλή η πρότασή σου. Εγώ τον κύριο Κρότσμαν εκπροσωπώ. Ευχαριστεί την Κρίστελ Σαλτελμόζε για τι συμβιβαστικέ τροπολογίες. Μπορεί να αποδεχθεί την 1 και την 7, αλλά υπήρχε και, υπήρχαν και αρκετέ τροπολογίε με τις οποίες δεν συμφωνεί και θεωρεί ότι χάνονται πολλές από τις δικές μας τροπολογίε, για παράδειγμα ευφυής, ε, κανονισμό ε, για σαφή διαχωρισμό μεταξύ του κανόνα για εναρμονισμένα και μη ε, εναρμονισμένα προϊόντα που μειώνουν το διοικητικό βάρος για του οικονομικού φορεί και επίσης δεν βλέπει τις τροπολογίες αυτές ε, να αντικατοπτρίζουν τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Ενδεχομένως να υπάρχει δουλειά ε, για σας κυρία Σαλδημόζη ακόμα. Το κοινοτικό σήμα τώρα και η υποχρέωση των οικονομικών φορέων να χρησιμοποιούν ε, τη σήμανση. Ο συνάδελφος ανησυχεί ότι αυτό θα δημιουργήσει μεγαλύτερη σύγχυση μεταξύ των ε, καταναλωτών αλλά και των επιχειρήσεων, γιατί η αρχή της πρόληψης που υποχρεούνται να επιβάλλουν οικονομικοί φορείς ε, σημαίνει με ασφάλεια, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι απολύτως βέβαιη η ύπαρξη αυτή. Η κοινοτική σήμανση, συμβιβαστική 4, πολλοί το θεωρούν ε, ότι είναι και σήμα ασφαλείας. Δεν ισχύει αυτό πάντα. Ως δικηγόρος όμως είσαι υπεύθυνο αν το χρησιμοποιήσεις εθελοντικά, αλλά άμα το χρησιμοποιήσεις ε, είσαι υπεύθυνο. Δηλαδή ε, το είδαμε αυτό με την περίπτωση κάποιων παιχνιδιών. Σε πολλές περιπτώσεις, για παράδειγμα, η κοινοτική σήμανση χρησιμοποιείται, αλλά πρέπει να υπάρχει και έλεγχος. Δηλαδή, σε μερικές περιπτώσεις, το ότι ελέγχεται από έναν παράλληλο οργανισμό σαν τον τούφ, για παράδειγμα, σημαίνει και ασφάλεια. Αν ελέγχεται ένα προϊόν που είναι ασφαλές και δίνει την κοινοτική σήμανση κανείς, τότε ε, η ευθύνη αφορά, καλύπτει και την ασφάλεια του προϊόντος. Πάλι συμφωνούμε. Τι ωραία. Αυτό που μου κάνει, που είναι δύσκολο να το επιτύχουμε, ε, σε μια συμφωνία έτσι γρήγορη, ίσως να πρέπει να προσπαθήσουμε όμως να το κάνουμε, τα ελκυστικά στα παιδιά προϊόντα. Θεωρεί ο συνάδελφος ότι είναι πολύ ευρύ, αυτό, αυτή, πολύ ευρύ αυτή η διατύπωση. Πρέπει δηλαδή να το διευκρινίσει κανείς. Η ιδέα πάντως καλή είναι. Όσον αφορά τις κυρώσεις, ε, πολλά υπόθηκαν για τις κυρώσεις. Ο κύριος Κρόιτσμαν ε, φρονεί ότι πρέπει να εναρμονίσουμε την, ε, τον κανονισμό σε όλα τα σημεία. Γιατί η εποπτεία της αγοράς καλύπτει όλα τα προϊόντα και το ίδιο θα έπρεπε να ισχύει, το ίδιο θα έπρεπε να ισχύει και στον κανονισμό αυτό. Επίσης, ζητά αξιολόγηση αντικτύπου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί είχαμε αποφασίσει κάτι τέτοιο στην Επιτροπή μας. Και να συνεχίσω τώρα στα Ολλανδικά. Γιατί θα μιλήσω για την τηλεόραση τη σχολική και είναι πιο απλό αν μιλήσω στα Ολλανδικά πρόεδρα εισηγητά. Ik wil graag nog wat zeggen over... Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για το Made in the EU σε ό,τι αφορά τη σήμανση για την κλωστοφαντουργία και το σχετικό φόρουμ. Ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ορίσει τους όρου με τους οποίους ε, μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει το Made in EU. Θα ήθελα να περιμένω πρωτού πούμε ότι α, το Συμβούλιο το θέλει το Made in the EU. Θεωρώ όμως ότι αν καταφέρουμε να το εισαγάγουμε θα μπορέσουμε να φέρουμε πολλές θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα σε άτομα υψηλής εξειδικευσής, τα οποία θέλουμε, τα οποία μπορούν να προσθέσουν κάτι συγκεκριμένο, απτό για τον καταναλωτή. Αν αγοράζω λοιπόν, ε, όταν αγοράζω μια γερμανική, ένα γερμανικό μηχάνημα και αναφέρεται ότι είναι made in Germany, ξέρω ότι αγοράζω ε, μηχάνημα υψηλής ποιότητας. Όταν αγοράζω δανέζικα τροφίμα, ξέρω ότι είναι ασφαλή. Έτσι λοιπόν, ε, όλοι έχουμε φυσικά τέτοιες εντυπώσεις για το marketing για το πώς μπορούμε να προαγάγουμε τα προϊόντα, πώς μπορούμε να προαγάγουμε στους καταναλωτές, πώς μπορούμε να διευκολύνει τον καταναλωτή όταν προέρχεται ένα προϊόν, για παράδειγμα, από, κάπου, από κάποια χώρα την οποία εμπιστεύομαι και στην Ευρώπη λοιπόν μπορεί να παράγουμε τέτοια ασφαλή προϊόντα. Θα πρέπει να θέσουμε όμως όρους για το πότε μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί το Made in Europe όταν ε, παρασκευάζεται για παράδειγμα και η συσκευασία μόνο. Όχι, θα πρέπει να γίνεται η σταρμολόγηση και η παραγωγή, η κατασκευή στην Ευρώπη. Τότε νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε το σήμα αυτό και αυτό θα είναι καλό και για το εμπιστοσύνη και για τον αγαπητή αλλά και για τον παραγωγό και για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε. Locking Garden, συνάδελφος, έχει το λόγο. Sorry, Chairman, I haven't asked for the floor. Συγγνώμη, εγώ δεν ζήτησα το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Η ομάδα σας όμως μας έδωσε το όνομά σας δεν είναι ότι εμείς το επινοήσαμε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Κρίμα που έφυγε ο προηγούμενος ομιλητής. Είναι σημαντικό, θεωρώ, να βρούμε μια συμβαστική λύση η οποία θα μας οδηγήσει σε μια λύση και με το Συμβούλιο, γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η πρόταση στην τρέχουσα θητεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το περιμένουμε 4-5 χρόνια τώρα. Και αυτό με απασχολεί βασικά και σε ό,τι αφορά το made in. Τι μπορούμε να κάνουμε για να πετύχουμε συμφωνία με το Συμβούλιο και πού το Συμβούλιο θα μπορούσε να τα ταχτυλώσει και πάλι. Δεν ενθουσιάζεται για το σύνολο της νομοθεσίας του Συμβούλιο, το ξέρουμε αυτό πολύ καλά. Δεν θέλω όμως για τον λόγο αυτό να κολλήσει το όλο ζήτημα στην ψηφοφορία. Θα ήθελα να περάσει στην τρέχουσα θητεία όπως σας είπα είναι λοιπόν ε, να κρατήσουμε μια γραμμή συμβιβαστική. Να ευχαριστήσω και τις δύο εισηγητρίες για τις προτάσεις τους και νομίζω ότι ε, σιγά σιγά μειώνουν το αριθμό των εκκρεμών ζητημάτων. Σε πολλά ζητήματα έχουμε προχωρήσει, υπάρχει μια καλή βάση η οποία φαίνεται και από τις ε, απαντήσεις των σκιωδών. Επίσης αυτό που ήταν σημαντικό στην έκθεση Μόζε σε ό,τι αφορά το C+, το σήμα αυτό. Όπως τα παρουσιάσατε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ περίπλοκα και δεν νομίζω ότι το Συμβούλιο υπάρχει περίπτωση να συμβιβαστεί. Αυτό που θεωρώ ότι είναι προβληματικό είναι ότι η πρότασή σας θα, όπως έχει η πρότασή σας, θα απέκλειε κάποιες μορφές ελέγχου, οι οποίες ήδη γίνονται στη Γερμανία. Δηλαδή θα δημιουργούνταν προβλήματα και σε χώρες όπου υπάρχουν σχετικές ε, προδιαγραφές. Το ερώτημα λοιπόν είναι ποια είναι η προστιθέμενη αξία για τον καταναλωτή και θα συμφωνήσω με τον κύριο Σφάμπε ότι εμείς στη Γερμανία κάναμε ελέγχου σε φυτεύματα, σε παιχνίδια, για παιδιά, σε τέτοια προβληματικά προϊόντα. ω τρίτη αξιολόγηση, άρα μια τρίτη πιστοποίηση, μάλλον μια πιστοποίηση από το τρίτο σώμα, δεν διασφαλίζει ότι τα προϊόντα δεν είναι ελαττωματικά. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να θεωρούνται υπεύθυνοι, υπέτοιοι και αυτοί οι φορείς τρίτης ε, πιστοποίησης. Στο σημείο 3 για παράδειγμα και στο σημείο 4 θεωρώ ότι είναι τελείως περιτά και το 2 θεωρώ ότι είναι περιτό. Έχω προβλήματα λοιπόν σε ό,τι αφορά το σήμαση, σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα του δικτύου ασφαλείας και εδώ θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Γιατί η καλύτερη νομοθεσία, το better legislation, τι σημαίνει ότι όταν κοιτάμε τομεακή νομοθεσία, θα πρέπει να διευκρινίζουμε σημαντικά ζητήματα άνεκ των υστέρων, χωρίς μελέτη αντικτύπου, χωρίς σχετική ακρόαση μέσω οριζόντιας νομοθεσίας. Ε, τίθεται ένα αμφιβόλο μια οριζόντια οδηγία, θεωρώ ότι είναι πολύ προβληματικό αυτό, όπως για παράδειγμα για τον κανονισμό για τα οικοδομικά προϊόντα. Γιατί ξέρετε δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ένα παράθυρο για παράδειγμα ε, ότι ένα παράθυρο είναι ασφαλέ. Το παράθυρο μπορεί να θεωρηθεί ασφαλέ μόνο εφόσον έχει τοποθετηθεί. Άρα τα οικοδομικά προϊόντα θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να εξισωστούν με άλλα προϊόντα. Και γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν τομιακέ νομοθεσίε και όχι οριζόντιε. Είναι πρόβλημα αυτό. Θα πρέπει να βρούμε μία λύση γι' αυτό. Είναι καλό αυτό που λέτε, ότι οι οικονομικοί διαχειριστές θα πρέπει να τηρούν τους όρους του New Legislative Framework, του νέου νομοθετικού πλαισίου. Αυτό το βλέπω και στις ε, συμβαστικές προτάσεις ε, της κυρίας Πιετικάινεν και τις δικές σας, ε, να είναι λίγο πιο απλή στη διατύπωση και να είναι να αφαιρθούν κάποια στοιχεία προβληματικά, για παράδειγμα το τι απαιτείται από τους καταναλωτέ, να τηρούν και να φιλάνε τις πληροφορίες της συσκευασία. Αυτό δεν βλέπω ότι έχει να κάνει με το New Legislative Framework. Δεν θα ήθελα να συμπεριληφθούν τέτοια στοιχεία. Νομίζω ότι ήταν πιο αποδεκτή η πρόταση χωρί τέτοια στοιχεία. Για την κυρία Πιετικά είναι τώρα. Καλό είναι ότι αναφέρεται το irrespective of the distribution channel, ανεξάρτητα από το κανάλι διανομή. γιατί δεν μιλάμε μόνο για offline και online. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν και άλλε μορφέ. Ε, πωλήσεων. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι σημαντική η ουδετερότητα σε ό,τι αφορά τον τρόπο πώληση. Εγώ θα ήθελα αυτό να μπει στο διδακτικό. Τώρα, αν συμπεριληφθεί κάπου αλλού, όπω είπαν οι σοσιαλδημοκράτε, αν συμπεριληφθεί στο συντολογικέ σκέψει, εντάξει, δεν έχω αντίρρηση, αλλά καλύτερα θεωρώ στο διδακτικό. Πιο μεγάλη νομική βεβαιότητα δίνει αυτό, θα το προτιμούσα σε ό,τι αφορά τι κυρώσει. Και στι δύο εκθέσει αναφέρεται καλό θα ήταν να διασαφινιστεί εξ αρχής. Με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια διατύπωση να ξεκαθαρίσει το θέμα. Να πω όμως και λόγια για τον κύριο Φόξ. Νομίζω ότι αναλωνόμαστε σε θέματα που είναι πολύ λεπτομέρειες και ψηλά γράμματα σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Και το κατά πόσο θα πετύχουμε τελικά μια πρόταση η οποία θα είναι better legislation δεν ξέρω. Γιατί εμείς θέλουμε το πλαίσιο να διευκρινίσουμε. Τώρα θα τις μεμονωμένε κυρώσει να το αποφασίσουν τα κάθε μελη Εμείς θα δούμε ένα γενικότερο πλαίσιο. Αν αποφασίσουμε επί κάποιων ε, μεμονωμένων, μετρημένων στα δάχτυλα βασικών στοιχείων, θεωρώ ότι θα ήταν πιο σωστό αυτό. Και έχω ανακοινώσει ήδη ότι θα αποσύρω τη σχετική μου πρόταση. Ευχαριστώ. Lockhart. Ευχαριστώ. Δεν πήρα το λόγο προηγουμένως, ε, γιατί ο συνάδελφός μου, ο καλός μου συνάδελφος Μάντες με προκάλεσε λιγάκι, γι' αυτό παίρνω το λόγο τελικά. Τέλος πάντων, ε, να το κάνω, να καταστήσω απολύτως σαφές, ε, ότι η άποψη των φιλελευθέρων δεν είναι αυτή που ανέφερε ο κύριος Μάντερς. Ξέρω ότι ο κύριος Μάντερς συμφωνεί πολύ με αυτή την ιδέα. Εμείς όχι. Εμείς πιστεύουμε ότι θα δημιουργούσε πολύ περισσότερο διοικητικό άχθος για τις ε, επιχειρήσεις ε, από τα προβλήματα που θα επέλυε. Οπότε να πω ε, για τα πρακτικά ότι δεν είναι αυτή η γενική γραμμή της ομάδος. Ναι και ευχαριστούμε. Κυρία Γκέπαρντ στη συνέχεια. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Να πω στον κύριο Λόκεγκαρτ ότι ήταν σαφές ότι ο κύριος Μάντελσον ο κύριος Μάντερς είπε αυτά που είπε Δεν μας παρουσίασε την άποψη της ομάδας του, ωστόσο αυτά που είπε συμφωνούν με την άποψη της δικής μου ομάδας και αυτό με χαροποιεί για τους δημοκράτες λοιπόν στο πλαίσιο αυτό το θέμα της προστασίας των καταναλωτών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα τρία σημεία θεωρώ ότι πρέπει να τονίσουμε. Πρώτον, η αρχή της πρόληψης. Πολύ σημαντική στην νομοθεσία αναφέρθηκε αυτό ήδη και θα θέλαμε να συνεχίσει να αναφέρεται. Ακόμα και αν έχει συμπεριληφθεί στο πρωτογενές δίκαιο. Και αυτό γιατί ενισχύεται η αρχή αυτή. Ξεκαθαρίζει το πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό για μας. Και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα παιχνίδια, προϊόντα και τα παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεύτερο θέμα. Το θέμα του CE+. Πολλές φορές το έχουμε συζητήσει και όντως, ακόμα και σε περίπτωση τρίτης πιστοποίησης, και πάλι, και πάλι μπορεί να υπάρχουν ανατοματικοί έλεγχοι. Αλλά, αν μέσω τρίτης πιστοποίησης και C+, του σήματος C+, διασφαλίσουμε ότι θα είναι λιγότερα τα προϊόντα τα οποία θα είναι αλληλεκτοματικά και θα ε, κινούνται στην αγορά, γιατί να μην το κάνουμε. Όχι επειδή δηλαδή έχουν γίνει σε κάποιες περιπτώσεις φάλματα να πούμε ότι «Α, εντάξει, θα αφήσουμε το σύστημα αυτό, γιατί έτσι κι αλλιώς γίνονται πάντα λάθη». Ε, δεν είναι δυνατόν αυτή την πολιτική να ακολουθούμε για τους καταναλωτές. Πρέπει να διασφαλίσουμε με το σήμα C+, να δημιουργηθεί μια προστιθέμενη αξία σε θέματα ασφάλειας. Γιατί το C το σήμα CE, το σκέτο, χωρίς το δεν είναι σύστημα, δεν είναι εγγύηση ποιότητα. Πολλοί καταναλωτέ το πιστεύουν όμω αυτό. Θα πρέπει να το διευκρινίσουμε. Είναι μόνο ένα σήμα το οποίο τη λέει ότι οι κανόνες που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν τηρηθεί. Τώρα ότι υπάρχει κόσμος που θεωρεί, μάλλον που παραποιεί αυτό το σήμα ε, το γνωρίζω. Δεν είναι αυτό όμως λόγος για να μην αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Αντιθέτως, θα πρέπει να κάνουμε καλύτερους ελέγχους σε ό,τι αφορά τη χρήση του σήματος. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι θα πρέπει να αποφύγουμε και να αφήσουμε τα, την τρίτη πιστοποίηση σε ό,τι αφορά το C+. Και θα δούμε, θα δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι πλειοψηφίες στην ομάδα μας στην Επιτροπή μας. Τώρα, για το σήμα προέλευσης. Πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Απασχολεί πολλούς πολίτες, γιατί θέλουν να ξέρουν που έχει παραχθεί, που έχει κατασκευαστεί το προϊόν. Και θέλουν να γνωρίζουν ότι το Made in EU, Made in Germany, France, Italy, όταν αναφέρεται, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και γι' αυτό λοιπόν αυτή η σήμανση, η προέλευση είναι πάρα πολύ σημαντική. Εγώ άλλες πληροφορίες έχω από αυτές του κυρίου Σφάπ. Ότι στο Συμβούλιο σε καμία περίπτωση δεν έχουν κατασταλάξει και ότι και στο Συμβούλιο είναι μεγάλη η απόσταση και η διάσταση των απόψεων και ότι καθόλου σίγουρο δεν είναι ότι θα καταψηφίσει το Συμβούλιο. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον Πολύ απλά να τα θέσουμε επιτάπητο στα θέματα αυτά, όπως τα πρότεινε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και να κάτσουμε να τα συζητήσουμε με το Συμβούλιο το τι είναι δυνατόν και τι δεν είναι δυνατόν και όχι των προτέρων να προτρέχουμε και να λέμε ότι α, κάποιος στο Συμβούλιο είπε ότι είμαστε κατά, άρα και εμείς ως Κοινοβούλιο θα είμαστε κατά. Όχι. Θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο συνειδητοποιημένοι, να θέσουμε το θέμα αυτό ως πολύ σημαντικό, ένα θέμα που ασχολεί τους πολίτες. Είμαστε λοιπόν εκπρόσωποι των λαών της Ευρώπης και όχι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων της Ευρώπης. Ευχαριστούμε και σας και τώρα κυρία Βάιλα. Ναι, και εγώ θα ήθελα να πω δύο λόγια για τα δύο αυτά σημεία. Καταρχάς για το C+. Νομίζω ότι σε μία αντικειμενική συζήτηση θα πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν μιλάμε μόνο για τη Γερμανία, μιλάμε και για 4-5 κράτη-μέλη μεγάλα, βιομηχανικά κράτη που έχουν παρόμοια σήματα. Δεν θυμάμαι τι έγινε ακριβώς πριν από 6-7 χρόνια στη σχετική συζήτηση, αλλά θυμόμαστε ότι αλλά αυτά τα σήματα εισήχθησαν από διάφορες επιχειρήσεις και όχι για την προστασία του καταναλωτή, αλλά από διάφορες επιχειρήσεις της ίδιας της βιομηχανίας, γιατί η βιομηχανία κατασκευής μηχανημάτων χρειάζεται τη σήμανση αυτή παρά το, το γεγονός ότι δεν απευθύνεται άμεσα στον καταναλωτή. Παρ' όλα αυτά, θυμάμαι όταν έγινε η πρώτη μεγάλη συζήτηση για την εποπτεία της αγοράς πριν από 6-7 χρόνια, ήταν και η κυρία Σαλτεμόζε, ο κύριος Λάμσντορφ, ο κυρία Ρούλε, αν δεν κάνω λάθος, είχα και εγώ, ήμουν και εγώ εισηγήτρια και όντω εισηγήτρια σε μια τέτοια έκθεση και τότε το Κοινοβούλιο αποφάσισε να καταργηθεί αυτό και στις ε, διαπραγματεύσεις για το Συμβούλιο πολέμησα εγώ προσωπικά να καταργηθεί μόνο αν περνούσε κάποια εναλλακτική λύση. Γιατί χωρίς κάποιο τέτοιο σήμα θα ήταν μοιραία η έκβαση για την βιομηχανία. Η βιομηχανία μαζί με την ε, επιστήμη λοιπόν, είχαμε πει τότε, θα έπρεπε να φτιάξει ένα πιο ποιοτικό σήμα. Αναρωτιέμαι λοιπόν τι έγινε τα τελευταία χρόνια, αν τα πράγματα είναι όπως με το Universal Charter και πει ο κλάδος ότι όσο δεν κάνει τίποτα η πολιτική δεν κάνουμε και εμείς τίποτα, αυτό πιστεύω ότι θα ήταν λάθος. Γι' αυτό λοιπόν στο πακέτο αυτό της ε, νομοθεσίας θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό ως πρόκληση. το σήμανση CE και η σήμανση η βιομηχανική. Αυτά θα πρέπει σίγουρα να συμπεριληφθούν. Τώρα το τι θα γίνει με το Συμβούλιο, ποια θα είναι η έκφαση, δεν μπορούμε αυτό να το προεξοφλήσουμε. Θα πρέπει να γίνουν διαπραγματεύσεις. Σε κάθε περίπτωση αυτό που είναι σωστό είναι η σήμανση C+, να θεωρηθεί μεταξύ, του σήματο. εσύ, Γιατί αν δεν συμβεί αυτό, πολύ απλά δεν θα συμβεί τίποτα τα επόμενα 6-7 χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν σίγουρα να κάνουμε ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για το made in. Να πω κάτι εντελώ διαφορετικό. Που σε, πολλά, σε πολλές χώρες προκαλεί μεγάλες αντιδράσεις και κυρίως στη Γερμανία. Νομίζω ότι ταξιδεύοντας τον κόσμο πηγαίνω και συχνά στην Ασία, βλέπω πολλά προϊόντα που αναφέρεται Made in the European Union, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρω όμως ότι προτρέχω. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται τα επόμενα δύο χρόνια και ως προς αυτό θα πρέπει με σαφήνεια να τοποθετηθούμε. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο τελευταίος ομιλητής, συνέλφος Στάιλερ, ή η κυρία Στάιλερ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα παίρνω το λόγο, αλλά μετά από κάποια σχόλια που άκουσα από συναδέλφου ε, που ε, είναι μέλη τη Επιτροπή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από μένα, θεώρησα ότι δεν είχα άλλη επιλογή. Όταν σχολιάζει το θέμα σε σχέση με τα εμφυτεύματα στήθους, για παράδειγμα, εγώ διάβασα το 2000 μία έκθεση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, τότε μιλούσαν με, για εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας, οι οποίες δεν είναι πολύ σημαντικές, ε, δεν θα πρέπει διεξοδικά να εξετάζονται κλπ. κλπ. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να λέμε ότι ειδικότερα για το θέμα των εμφυτευμάτων στήθους, αν οι συστάσεις είχαν ληφθεί υπόψη, δεν θα είχαμε φτάσει στην κατάσταση που αντιμετωπίσαμε και που αντιμετωπίζουν πολλές ε, εκλογικές μα περιφέρειες, δεν ξέρουν ακριβώς τι υπάρχει μέσα στο σώμα τους. Δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε αυτό το θέμα, γιατί είναι ένα θέμα εγκληματικής ε, αμέλειας ε, και απάτης. Πρέπει να πούμε ότι ορισμένα, σε μερικέ περιπτώσεις εγκληματικότητα και απάτη δεν δεχόμαστε σε τέτοια πράγματα. Ίσως ορισμένα δηλαδή συγκεκριμένα ε, σημεία και θέματα να, έπρεπε, να τα πρέπει όντω να τα ονομάσουμε. Όσον αφορά τώρα το θέμα που ανέφερε κάποιος από τους συναδέλφους, μου έκανε πολύ εντύπωση αυτό το είδος κανονισμού, ως ιδέα έχει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σύνολο κανόνων που ισχύουν για όλα τα κράτη-μέλη, θα πρέπει να είναι απλή και σαφής και όταν πηγαίνουμε στις διαπραγματεύσεις ξέρουμε ότι αυτή είναι η χρονική στιγμή που ε, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το περίπλοκο που έχουμε μπροστά μας και θα ήθελα πραγματικά να επενέσω τη συνάδελφο για τη δουλειά της. Δεν είναι καθόλου εύκολο όταν οι συνάδελφοι μιλούν για τις διαπραγματεύσεις δεν θα έπρεπε να, υπο, να υποτιμούν το πολύπλοκο και τη δυσκολία των διαπραγματεύσεων, αλλά ε, πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό είναι τμήμα της δουλειάς μας και κρίμα που έφυγαν οι συνάδελφοι, θα πρέπει να έχουν μείνει εδώ να το συζητήσουμε. Θα ψηφίσουμε την Πέμπτη, έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας, αλλά καθόμαστε γύρω-γύρω από το τραπέζι όλοι και συζητάμε και οι συνάδελφοι που θα έπρεπε να προσπαθούν όσο το δυνατόν περισσότερο να λύσουν ε, μαζί με εμά τα προβλήματα, να εξασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα που υπάρχουν στην αγορά είναι ασφαλή και ότι αυτά τα οποία αγοράζουμε, αυτά που έχουμε, έχουν τη σωστή ετικέτα που εγγυάται την ασφάλεια των προϊόντων. Υπάρχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά υπάρχουν και οι καταναλωτές που αγοράζουν τα προϊόντα των επιχειρήσεων αυτών. Οπότε θα ήθελα να ευχαριστήσω και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στη συνάδελφο για τις διαπραγματεύσεις. Ελπίζω να καταλήξουμε σε κάτι το οποίο πραγματικά θα μας ε, βοηθήσει όλους και θα είναι προφελές για όλους. Ο κύριος Λόκεγκάρτ. Ναι, μάλλον με τιμωρούν επειδή άργησα. Θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα εκ μέρους του συναδέλφου Χέλτικ. Θα ήθελε να ζητήσει συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Θα ήθελε επίσης να ευχαριστήσει την εισηγήτρια για τη δουλειά της, όπως και για τις συμβιβαστικές τροπολογίες που ε, διατύπωσε. Ε, το πεδίο εφαρμογής, ε, η διάκριση μεταξύ των ασύμβατων προϊόντων, κίνδυνος των προϊόντων, εφαρμογή των, της τη αγοράς, όπως επίσης και η θέση των οικονομικών φορέων είναι ικανοποιητικές σχετικές τροπολογίες, όμως υπάρχουν ορισμένα ζητήματα όπως οι κυρώσει, για παράδειγμα που θα έπρεπε κατά τη γνώμη του να επιβάλλονται για κάθε περίπτωση ακόμη και αν ε, η παράβαση ε, είναι ε, κατόπιν αμελίας, δεν είναι θελοντική δηλαδή, είναι ακούσια. Ε, Παρ' όλα αυτά είναι κάτι το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη. Πρέπει να είναι αποτρεπτικό ο χαρακτήρα, αλλά και ανάλογο ο χαρακτήρας των κυρώσεων Όσον αφορά την αρχή της πρόληψης, ε, είναι μια γενική αρχή της συνθήκης. Ο κύριος Γιαλούτη θα μπορούσε να υποστηρίξει την αναφορά στο άρθρο 1 που λέει ότι ο κανονισμός ε, ορίζει ένα πλαίσιο που συνάδει με την αρχή της πρόληψης. Όσον αφορά τα εκκρεμή ζητήματα άλλων συμβιβαστικών ε, τροπολογιών, θεωρεί ότι είναι τεχνικά και ελπίζει ότι αύριο στη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών θα επιληθούν. Ευχαριστώ. <clears throat> Και τώρα, η κυρία Σπάν έχει το λόγο από πλευρά Επίτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και όλου του βουλευτέ, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ ωφέλιμο το ότι ακούμε τα τις απόψεις σας ε, σήμερα. Δεν θα σας απασχολήσω πολύ, να σας δώσω κάποιες διευκρινήσεις γιατί φτάνουμε σε ένα κρίσιμο σημείο στο πακέτο αυτό. Καταρχάς, θα θέλαμε να καλωσορίσουμε τις τροπολογίες που κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, που διευκρινίζουν κάποιους ορισμούς όπως ε, ε, για παράδειγμα, του ευάλωτου καταναλωτέ, τα προϊόντα που απευθύνονται στα παιδιά, θα πρέπει οι προτάσει μα να είναι σαφεί. Για την αρχή τη πρόληψη, είπαμε και στο παρελθόν ότι για μα πρόκειται για μια αρχή του νόμου που εφαρμόζονται κατά το δέοντα τρόπο. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει κάποια, α, κάποια θέματα στο Συμβούλιο. Αυτό το επαφίουμε στον νομοθέτη για τα πια, πιο δύσκολα θέματα τώρα. Το C+ η σήμανση C+. Χαιρόμαστε για τα σημερινά σχόλια γιατί βοηθούν να καταλάβουμε την πρόταση αυτή. Θα θέλαμε να επενθυμίσουμε εδώ σε όλους ότι αυτή η πρακτική για το σήμα CE είναι καλά εντρεωμένη. Παρ' όλα αυτά δεν προορίζεται ως σήμα ασφάλειας, αλλά όλα τα προϊόντα τα οποία κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά, στην ενιαία αγορά, υποτίθεται ότι είναι ασφαλή. Άρα ορισμού όλα τα προϊόντα με τη σήμανση CE είναι ασφαλή. Αυτό που είναι σημαντικό είναι το εξή. Αν ποτέ εξετάσουμε την ιδέα ενό συστήματο, θα πρέπει να είναι ένα σύστημα λειτουργικό με σαφή κριτήρια και δεν είμαι βέβαιη ότι έχουμε κατανοήσει ακόμη το πώς θα εφαρμόζονταν στην πράξη ένα τέτοιο σύστημα και πώς δεν θα προκαλούσε σύγχυση με το ίδιο υφιστάμενο σήμα CE και σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές και τους ε, διαχειριστές θα είχαν δηλαδή δύο κατηγορίες προϊόντων στο μυαλό τους. Αυτά λοιπόν είναι ερωτηματικά που θέλω να θέσω προς τους ε, βουλευτές για τις κυρώσεις. Είδαμε κάποιες ενδιαφέρουσες ιδέες Μία έκκληση, μία έκκληση σας απευθύνω, επιτρέψτε μου, να εξετάσουμε τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις οποίες μπορούμε να ασκήσουμε. Δεν είμαι βέβαιη κατά πόσο από νομική άποψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε θέση να, δημιουργηθεί, να δημιουργήσει μαύρες λίστες, να διαχειριστεί ένα σύστημα το, όπως προτείνεται στην παρούσα φάση για το ηλεκτρονικό εμπόριο να ξεκαθαρίσω ότι ναι, όντως η ιδέα είναι η πρόταση να ισχύει και online και offline και οι έλεγχοι αφορούν και τα ψηφιακά προϊόντα και σκοπός μας είναι όταν θα έρθει η μαγική στιγμή ε, υιοθέτηση των προτάσεων να δώσουμε κατευθυντήριες γραμμές για το πώς η νομοθεσία αυτή θα ισχύσει στον ψηφιακό κόσμο. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη πρόκληση. Χρειαζόμαστε κατευθυντήριες γραμμές από εμπειρογνώμονες. Τέλος, σε ό,τι αφορά το θέμα της χώρας προέλευσης, είναι πολύ σημαντική η συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να σας υπενθυμίσω γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε αυτή τη σήμανση της προέλευσης. Θέματα εμ, 10% των προϊόντων μας είναι άγνωσης προέλευσης, ανίχνευσης. Αν μπορούμε λοιπόν αυτό το 10% να το διορθώσουμε, γιατί όχι. Κατά δεύτερον, πρόκειται για μια υφιστάμενη πρακτική σε πολλά κράτη-μέλη, από πολλού παραγωγού. Και σε πολλέ δικαιοδοσίε υφίσταται αυτή η πρακτική. Λοιπόν, αν το κάνουν αυτό οι έμποροι, γιατί να μην το κάνουμε κι εμεί αυτό. Και όπω είπαν πάρα πολλοί βουλευτέ στην πράξη αυτό είναι κάτι που είτε γίνεται. Εκ παραλίλου, να σα πω ότι είδαμε τροπολογίε από άλλε επιτροπέ εδώ του Κοινοβουλίου, που κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση από τη διαγραφή του όρου αυτού μέχρι και τη βελτίωση προκειμένου να παράδειγμα πρόταση η οποία λέει να είναι ανοιχνεύσιμη ανοιχνεύσιμα όλα τα συστατικά ενός προϊόντος. Νομίζω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η πιο ρεαλιστική. Τέλος, για μένα το πιο σημαντικό που άκουσα σήμερα ήταν το θέμα της έκκλησης για το χρονοδιάγραμμα έχει φτάσει το πλήρωμα του χρόνου. Είναι όριμη η χρονική στιγμή. Και σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο, σε ό,τι αφορά το θέμα της αγοράς προέλευσης, έγινε συζήτηση στον Κορεπέρ και υπάρχει προθυμία λοιπόν να εξευρεθούν λύσεις στον τομέα αυτό. Βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα σε μία φάση όπου το θεσμικό όργανο αυτό είναι δεσμευμένο χαιρόμαστε. Θα σας υποστηρίξουμε στην ε, ε, υιοθέτηση του πακέτου αυτού στην τρέχουσα θετία του Κοινοβουλίου. Θεωρούμε ότι αποτελεί αυτό καθήκον μας προς τους πολίτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Σύμφωνα με τη μερισία διάταξη θα δώσουμε το λόγο στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχά, συνάδελφοι, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ καλά και χρήσιμα σχόλιά σας. Νομίζω ότι θα γίνουν κάποιες διαπραγματευτικές συνεδριάσεις ε, ακόμα πριν ε, ε, ψηφίσουμε την Πέμπτη. Όμως θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα για το C+. Να πω το είπα και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Αν εγώ αποφάσιζα, πιστεύω ότι την κοινοτική σήμανση θα έπρεπε να την έχουμε μόνο στους τεχνικούς φακέλους που έχουν να κάνουν με τα προϊόντα και όχι πάνω στα προϊόντα, γιατί είναι παραπλανητικά για τους καταναλωτές. Αλλά η εποπτεία της αγοράς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έμαθα ότι προτιμούν η σήμανση να υπάρχει πάνω στα προϊόντα και γι' αυτό ακριβώς λέω ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να λαμβάνουν λίγο με καλύτερη ενημέρωση που θα μπορούσε να προσθέτει κάτι σε αυτό. Γι' αυτό πρότεινα C+, κάτι το οποίο θα μπορούσε να συνδέεται με όλα τα προγράμματα που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, το γερμανικό DS. Θα μπορούσε να έχει και εσύ plus δίπλα. Ε, είναι προαιρετικό, μπορεί να χρησιμοποιείται και σε μη αρμονισμένα προϊόντα. οι ανεξάρτητοι δοκιμαστές ε, θα έπρεπε να είναι αξιόπιστοι στο αποτέλεσμα ως το προς το πόρημά τους, ώστε αν κάποιο, κάποιο προϊόν δεν είναι ασφαλές να μπορούν να μηνύσουν οι καταναλωτές. Δεν θέλω να το συζητήσουμε, απλώς θέλω να το εξηγήσω λιγάκι, να το αποσαφηνίσω. Όσον αφορά το ε, κατασκευάζεται στην τάδε χώρα, το made in, θα σας πω ένα πράγμα. Αν δει κανείς πίσω από το iPhone του, θα δει ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη ένα made in. Λέει για παράδειγμα ότι έχει σχεδιαστεί στην Καλιφόρνια, αλλά έχει συναρμολογηθεί στην Κίνα. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες ε, ήδη εξάγουν στη ΣΥΠΑ και πρέπει να συμμορφώνονται με τον κανονισμό αυτό. Αν θα μπορούσαμε να ευθυγραμμίσουμε κάπως τις ιδέες μας εδώ στην Ευρώπη με τις ε, υποχρεώσεις ε, που υπάρχουν στις Ηνωμένε Πολιτείε, δεν θα ήταν επιπλέον βάρος, ε, θα ήταν βοήθεια προς τις επιχειρήσεις. Αυτό θα μπορούσε να είναι κάποιο είδου συμβιβασμό που θα μπορούσαμε να εξεύρουμε όταν θα πηγαίνουμε να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο, εμείς ως Κοινοβούλιο. Και τέλος, ένα ακόμη σχόλιο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγγνώμη που θα το επαναλάβω, το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι βοηθάει πολύ όταν κάθεται κάποιος εδώ στην Επιτροπή μας λέτε ποια είναι, ποιος είναι ο σωστός τρόπος ε, να κάνουμε τα πράγματα. Καλύτερα τα αφήσω στους νομοθέτες. Είναι ο καλύτερος τρόπος να βρούμε τη λύση. Μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι θα θέλατε να μην αλλάξουμε τίποτα πολύ στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εμείς δεν δουλεύουμε έτσι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε ίσως καλύτερα να μην σχολιάζετε τις άμεσες διαπραγματεύσεις που λαμβάνουν χώρα εδώ στις, ε, στη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρω ότι θέλετε να μας βοηθήσετε, αλλά στην ουσία δεν μας βοηθάτε. Καλύτερα να τα αφήσετε στους ευρωβουλευτές, να καταλήξουν στην θέση του Κοινοβουλίου και είμαι πεπισμένη ότι μπορούμε να βρούμε καλές λύσεις. Θα έχουμε συναντήσεις ε, πριν από την Πέμπτη και την Πέμπτη θα ψηφίσουμε και είμαι αισιόδοξη ως προς το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ για τα πολύ καλά και χρήσιμα σχόλιά σας. Σας ευχαριστούμε. Ο συνάδελφος Σφάμπ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά Μίλησα για την έκθεση εξ ονόματος της κυρίας Ρόιτοβα. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω πρόβλημα να ψηφίσουμε, αλλά θέλω να ψηφίσουμε για ουσιαστικά θέματα. Δεν θέλουμε να προσπαθήσουμε να βρούμε την πλειοψηφία του Συμβουλίου, αλλά καλό θα είναι να συμμετέχει και η Επιτροπή μας και όχι απλά να το αφήσουμε αυτό σε κάποιους συναδέλφους στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι καλό είναι να συζητήσουμε εδώ πολιτικά. Να μην ε, απορρίψουμε εξ αρχής κάποιες ιδέες. Καταρχάς, ε, είπα ότι δεν έγινε μελέτη δικτύπου για το άρθρο 7. Δεν εξηγείται πώς υπολογίζονται τέτοια συστήματα. Δεν υπάρχει λοιπόν impact assessment. Η κυρία Σάλτε Μόζε μίλησε δικαίως για το Made in USA σωστό και ενδιαφέρον, αλλά οι κανόνες αυτοί δεν έχουν να κάνουν με τον τελωνιακό κώδικα. Αλλά αυτό ισχύει στη δική μας περίπτωση. Γι' αυτό λοιπόν σας ερωτώ, γιατί λειτουργούν αυτά στη ΣΥΠΑ και γι' αυτό δεν λειτουργούν σε εμά τα πράγματα στον τελωνιακό κώδικα. Δεν υπάρχει αληθοφανής, ε, μάλλον ε, σωστή αποτύπωση για το πού ε, παράγονται τα προϊόντα Για παράδειγμα, μπορεί κάποιο προϊόν να παράγεται στον Καναδά, αλλά να έχει έξω από την Ιταλία. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Όταν κάποιος λέει made in Italy, made in Germany, προσπαθεί να δημιουργήσει την εντύπωση ότι εκεί παράγεται το προϊόν. Και οι ανταγωνιστές ζητούν να ισχύει αυτό, να υπάρχει εναρμόνιση, σύμφωνη, αλλά σωστή εναρμόνιση και να μην επικεντρωνόμαστε στην τελευταία, στον τελευταία χώρα παρασκευή. μόνο. Αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζω. Αλλά θα δούμε τι θα γίνει και στην ψηφοφορία αύριο. Ολοκληρώσαμε έτσι. Παρακαλώ. Η ε, κυρία Κέπχαρτε. Αγαπητέ συνάδελφε, πάμε λίγο πιο μεγάλη συνοχή να μα έχετε. Πριν μα λέγατε από το Συμβούλιο, αποφάσισε ότι το άρθρο 7 πρέπει να φύγει και μας ε, προτείνεται να το καταργήσουμε. Τι να συζητήσουμε τότε στο Συμβούλιο, μα συγγνώμη κιόλα. Είτε το ένα ισχύει είτε το άλλο. Δεν μπορείτε να μας λέτε ότι επειδή ο νομοθέτης, μάλλον να λέει και δύο νομοθέτες να διαγραφεί το θέμα αυτό και μετά να το συζητήσουμε αν θα προσταθεί ή όχι, μα δεν θα γίνει συζήτηση μετά. Και νομίζω ότι ακριβώς το θέμα αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό θα πρέπει να το συζητήσουμε και με το Συμβούλιο. Και γι' αυτό είμαι υπέρ. Γιατί δεν ξέρουμε τι συζητιέται στο Συμβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να τηρηθεί το άρθρο 7 εδώ προκειμένου να έχουμε και μια βάση για τη συζήτηση. Γιατί αν δεν υπάρχει καμία βάση, ε, να τα μαζέψουμε να φύγουμε. Σα ευχαριστώ Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους οι οποίοι πήραν τον λόγο. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε το θέμα και πάμε στο σημείο 10 τώρα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μπάστος. Πώς. Ναι, εντάξει. Την κυρία Μπάστος την ε, περιμέναμε. Va bene, riprendiamo. La signora Bastos è arrivata. η κυρία Μπάστος. Γι' αυτό να δούμε το 4 και 5. Μάλλον να πάμε τώρα στο επόμενο. για το marketing Κυρία Μπάστος είναι εδώ. Μισό λεπτό. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κάποιος θόρυβος υπάρχει εδώ μέσα και δυσκολεύομαι να ξεκινήσω. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Παρακαλώ όποιος επιθυμεί να συζητήσει μήπως θα μπορούσε να αποχωρήσει και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Το απόγευμά μου σήμερα ήταν πραγματικά δύσκολο. Και ζήτησα από τον Λεσμίτ ε, να αλλάξει μαζί μου για την παρουσίαση και θα έπρεπε να δούμε να ψηφίσουμε στην Επιτροπή Γυναικών ε, μια σημαντική έκθεση και μετά να είμαι και εδώ για να δούμε τις τροπολογίες. Σε ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για αυτές τις τροπολογίες που υπέβαλαν για τα δύο κείμενα. Και εγώ σαν εισηγήτρια έχω τις δικές μου τις τροπολογίες που θα ήθελα να προτείνω για το κινητικό σήμα για την ε, οδηγία για τα σήματα, τα κοινοτικά σήματα κοινοτικό σήμα και αυτά τα 27 αφορούν την ελευθερία έκφρασης, την συγκριτική διαφήμιση, τα όσα αιτιολούν μια άρνηση και δεν θα ήταν ε, εύκολο να βρούμε ένα όρο για τα 15 και 16 σε σχετικά με το αρχικό της γνωμοδοτήσης μου και επίσης και άλλες ε, τροπολογίες για την προέλευση του προϊόντος όπως επίσης και την ε, online, τον online έλεγχο. Ίσως από τις τροπολογίες είναι το πιο λεπτό θέμα με, όπου συμφωνούν οι λιγότεροι συνάδελφοι. Θα μπορούσα να συζητήσω μαζί τους για να δούμε πώς θα ξεπεράσουμε αυτές τις διαφορές μας. Προσπαθούμε να πετύχουμε μια σύγκληση. Προσπαθούμε να πετύχουμε ένα κοινό παρανομαστή. Και στις νομοδοτήσεις τότε είχα πει εγώ ότι δεν χρειαζόταν να διατυπώσουμε τα πάντα τις σημερινές του συστήματος. Δεν θα πρέπει να επιφέρουμε εκεί μια επανάσταση γιατί αποτελούν βάσεις που έχουν πάντα μια αξία. Τι θα επιθυμούσαμε είναι να δώσουμε μια συνέχεια στις νομοδοτήσεις με αυτές τις τροπολογίες και θέλουμε να απλουστεύσουμε την όλη διαδικασία για το κοινοτικό σήμα και να μην ε, κοστίζει και τόσο ακριβά. Α, λοιπόν, ε, Δύσκολο πάντως για μια συμφωνία μεταξύ μας και γι' αυτό θα ήθελα να έρθω σε επαφή με τους συναδέλφους με αυτό το στόχο. Να εξηγήσω τώρα μία τροπολογία που υπέβαλα εγώ και είναι το, το 25 του 9 άρθρου και το άρθρο 14 επίσης. Το κείμενο της Επιτροπής τι λέει ότι για ένα κοινοτικό σου σήμα θα μπορούσε βάσει αυτού να απαγορευθεί και η εισαγωγή προϊόντων σύμφωνα με το 3C. Και όσον αφορά την αποστολή αυτού του προϊόντος που έχει εμπορικό χαρακτήρα, εγώ θα ήθελα να προτείνω το εξής. Θα ήθελα να αλλάξουμε την πρόταση και θα θέλω να πούμε και παρακαλώ προσέξτε ο κάτοχος ενός σημαντικού σήματος θα μπορούσε να αποτρέψει με τη βοήθεια του κράτους του εθ, της χώρας την εισαγωγή εμπορευμάτων ε, σύμφωνα με το άρθρο 3C και την προσφορά προϊόντων σύμφωνα με το 3Β και ο αποστολέας ή ε, διάμεσος ε, που να γίνεται κάτι online και ένα που έχει εμπορικό στόχο. Εδώ συμπεριλαμβάνουν λοιπόν και το εμπόριο online που συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την πρότασή μου για την μετατροπή. Ο στόχος λοιπόν ποιος είναι. Θα ήθελα ο κάτοχος αυτού του εμπορικού σήματος καθώς και από πλευράς ε, χώρας να μπορούσαν να αποτρέψουν την εισαγωγή προϊόντων ή επίσης παράνομων απομιμήσεων και σε όλους όσους ενέχονται στην ενέργεια αυτή, τον Αποστολέα, τον ένα τον άλλο και από τη στιγμή που έχουμε μια online συναλλαγή, από τη στιγμή που έχει εμπορικό στόχο να απαγορεύσουμε στον Αποστολέα και στον ενδιάμεσο αν υπάρχει ένας εισαγωγέας που τα καταφέρει και κάνει εισαγωγή προϊόντων. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εμείς θα πρέπει να τον ρωτηθούμε, θα πρέπει να έχουμε μια απάντηση. Ξέρουμε ότι η απομίμηση αποτελεί ένα εμπόδιο γιατί καταστρέφει θέσεις εργασίας. Μιμείτε το αρχικό προϊόν. Είναι εις βάρος της ευρωπαϊκής οικονομίας και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο επίσης την ασφάλεια και την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Γι' αυτό θα πρέπει αμέσως να αντιδράσουμε θαραλέα μάλιστα. Και ακόμη, έχουμε και στοιχεία εκατομμύρια απομιμήσεις που κατασχέθηκαν 115 εκατομμύρια από το 2011 που κατασχέθηκαν. Η αξία τους είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2011 είναι και δυνητικά επικίνδυνα προϊόντα για την υγεία των καταναλωτών. Θα πρέπει λοιπόν να τα πολεμήσουμε γενικότερα. Και να δούμε τι γίνεται επίσης με τα δικαιώματα. Ε, ας πούμε ότι κάποιος θέλει στο YouTube να φέρει ένα βίντεο και αυτό το βίντεο όμως αποσύρθηκε για παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων. Εδώ το ίδιο για ένα καταγεγραμμένο εμπορικό σήμα και από τη στιγμή που ξέρουμε ότι υπάρχει μια σχετική πλατφόρμα θα πρέπει να δούμε και ο κατόχος αυτού σήματος και το εθνικό κράτος θα μπορέσουν να ζητήσουν από αυτήν την πλατφόρμα να, από αυτό το μέσο να αποσύρει τα προϊόντα από την αγορά γιατί είναι απομιμήσεις παράνομες. Αυτό. Απλό μπορώ να σας δώσω και παραδείγματα αν δυσκολεύεστε να το καταλάβετε, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το σαφές και συγκεκριμένο, μπορούμε έτσι να διευκρινίσουμε τη θέση μας σχετικά. Και επίσης υποφελούμε για να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν ξέρω βέβαια αν είναι παρόν κάποιος εκπρόσωπος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι κάποιος εδώ? Όχι. Κανείς. Εντάξει, αργότερα τότε. Παρακαλώ τους συναδέλφους να μου πούν ποια είναι η απόψή τους σχετικά με τις παρατηρήσεις για αυτά τα στοιχεία και ευχαριστώ ακόμα μια φορά όλους σας και αναφέρομαι στους συναδέλφους οι οποίοι υπέβαλαν, κατέθεσαν τροπολογίες σχετικά. Σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Κυρία Γκέφχαρτ, ε, παρακαλώ μήπως επιθυμείτε να λάβετε το λόγο, όχι. Τότε, Κρότσμαν, ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την συνάδελφο Μπάστος για την πολύ καλή έκθεση. Κάποιες προσθήκες στην τροπολογία μου προσπάθησα να διευκρινίσω και να φτιάξω πιο ελκυστικό, ελκυστική την διαδικασία σε ό,τι αφορά και τη βιωσιμότητα ε, ε, του συστήματος προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά τα θέματα των τελών και των προθεσμιών. Εγώ λέω να τηρηθούν αυτές οι προθεσμίες, οι οποίες έχουν ε, αποδειχθεί ότι λειτουργούν. Να μην δυσκολέψουμε λοιπόν τα επιχειρήσεις και σε ό,τι αφορά θέματα διαμεσολάβησης εξώδικών αποφάσεων. Θα πρέπει πριν από την αρχή της επίσημης διαδικασίας, της επίσημης αγωγής να χρησιμοποιούν αυτά τα μέτρα και να διατύφονται σχετικέ πληροφορίες. Να υπάρχει σωστή πιστοποίηση προκειμένου να ξέρουν ε, τα μέρη ποιες δυνατότητες έχουν επίσης στην ευρωπαϊκή αγορά να υπάρχει ένα κράτος μέλος ή μια περιφέρεια της, ε, του κράτους μέλους να προστατεύουν τα προϊόντα αυτά. Με πράξεις ε, κατά εφαρμογή να μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει τέτοιες δράσεις και να επενδύει σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων προκειμένου να μην φεύγουν όλα αυτά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο έλεγχος λοιπόν των προτάσεων αυτών θα πρέπει να γίνει και στο μέλλον να γίνεται από τις εθνικές αρμόδιες υπηρεσίες χωρίς όμως ε, αυτόματα διαδικασία σε ό,τι αφορά τις αιτήσει αυτές. Υποστηρίζουμε τις πιο πολλές προτάσεις των συναδέλφων. Θα πρέπει οι προτάσεις Παντσέρη για την χρήση ενός σήματος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει ως τώρα αμφιβολία για τη σήμα προέλευσης σε ό,τι αφορά και τη χρήση στο ίντερνετ. Και στην τελευταία συνεδρίαση τόνισα ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την υποστηρίζω σε ό,τι αφορά τα εθνικά αυτά συστήματα. Αυτό ισχύει σε περιπτώσεις που είναι ενδιάμεσο σταθμός η Ευρωπαϊκή Ένωση για άλλα κράτη σε ό,τι αφορά τα παραποιημένα αυτά προϊόντα τα οποία οι πολίτες, οι καταναλωτές μπορούν να παραγγείλουν από το διαδίκτυο. Αυτό θεωρούμε όμως δεν θα πρέπει να ισχύει όπως η κυρία Μπάστος και μεταξύ των ιδιωτών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κάποιος άλλος? Όχι. Ο σκιώδης ηγητής, Επιτροπή, μήπως κάποιος από την Επιτροπή θα επιθυμούσε να λάβει το λόγο. Ecco, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πολύ καλά. Είναι παρόν εκπρόσωπος της Επιτροπής. Άρα λοιπόν απευθύνω το ερώτημα. Ποια είναι η άποψή τους ε, για τους αποστολείς. Εκεί είμαι πως θα συμμετάσχουν κι άλλοι και τη βάση online για τη δυνατότητα δηλαδή κάποιου ελέγχου και καταγγελίας σε περίπτωση πλαστών απομιμήσεων και σε περίπτωση κατάσχεσης μετά από καταγγελία αυτών των προϊόντων. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Τι κάνουμε. Παρακαλώ. Η άποψη της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής ποια είναι. Να πω ότι ευχολώ ε, ότι ευχαριστώ τον κύριο Κρόιτσμαν για αυτές τις τροπολογίες, τις λογικές, τις ε, ιδιαίτερα χρήσιμες που κατέθεσε στις ε, δύο αυτές νομοδετήσεις και να δούμε και για το τι καλύτερο μπορεί να γίνει για τον εξωτερικό μεσολαβητή και τα υπόλοιπα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια δυσκολία, μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος ο πρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη που άργησα. Παράλληλες συζητήσεις ε, ε, γίνονται και στην ε, Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και γι' αυτό δεν μπορούσα να έρθω νωρίτερα. Δύο γενικά σχόλια θα ήθελα να κάνω σε σχέση με συγκεκριμένες τροπολογίες. Θα προσπαθήσουμε επίσης να απαντήσουμε στα ερωτήματα που θέτει η συγγήτρια. Δύο ανησυχίες έχουμε όταν βλέπουμε τις τροπολογίες. Πρώτη, τροπολογίες ε, η 26 για την αναδιατύπωση της οδηγίας και τροπολογία 31 για την αναδιατύπωση του κανονισμού του κοινοτικού σήματος. Αυτή τη στιγμή το νομικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει μία, ένα καθεστώς ε, εκπνοής Αυτό το καθεστώ όμω δεν είναι τμήμα των προτάσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής, οπότε μα κάνει λίγη εντύπωση το ότι είδαμε ότι υπήρξαν τροπολογίες παρόλα αυτά και για τις δύο διατάσεις, ε, οι οποίες ε, δεν ε, αφορούν προτάσεις που προήλθαν από μας και κάτι ακόμη. Θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολήθηκε πάρα πολύ μέσω μιας περιεκτικής μελέτης της δεκαετίας του 90 όπως επίσης και διαβουλεύσει με τους εμπλεκόμενους φορείς, πιστεύουμε ότι επί τη βάση των πορίσματων αυτών, των πορίσματων αυτών δεν θα ήταν ε, καλή ιδέα να αλλάξει το τρέχον καθεστώς. Δεν βλέπουμε όμω αποδεικτικά στοιχεία ότι κάτι τέτοιο θα ε, μείωνε τις τιμές καταναλωτή μακροπρόθεσμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα επίσης να πω ότι η πρόσφατη περιεκτική μας αξιολόγηση για τη λειτουργία του συστήματος κοινοτικού σήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν μια μελέτη από το Ινστιτούτο Max Planck ε, κάτι το οποίο έδειξε ότι δεν υπήρξαν επιβλαβείς συνέπειες του υπάρχοντος καθεστώτος ε, ούτε έχει σχολιαστεί από άλλες ενώσεις καταναλωτών ή εμπλεκόμενους φορείς κατά τη διάρκεια της μελέτης. Ένα δεύτερο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω και είναι κάτι το οποίο έχω τονίσει και στην παρέμβασή μου στις προηγούμενες συνεδριάσεις είναι η μεγάλη σημασία που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πιο αποτελεσματικά μέσα αντιμετώπισης ε, ε, των παραποιημένων προϊόντων και του διεθνούς εμπορίου αυτών Θέλουμε μία απλή και αποτελεσματική λύση για τα υποδιαμετακόμιση προϊόντα. Δεν θέλουμε τέτοιου είδους προϊόντα παραποιημένα να απολούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θέλουμε και να αποφύγουμε η Ένωση να αποτελήσει ένα, ένα κέντρο παγκόσμιας ε, διανομής αυτών των προϊόντων. Για τα ερωτήματα τώρα της εισηγήτριας νομίζω ότι έχουν να κάνουν ε, με την πρόταση που κάνουμε σε σχέση με το άρθρο 10 παράγραφος 4 της ε, ε, οδηγίας και το άρθρο 9 παράγραφος 5 όσον αφορά τα εμπορικά φορτία που αποστέλλονται ε, σε ιδιώτες από το εξωτερικό. Το ερώτημα είναι κατά πόσο θα πρέπει αυτό να συμπληρωθεί αν δω την τροπολογία 25 που αναφέρεται όχι μόνο στα φορτία, αλλά και σε άλλους ενδιάμεσους φορείς. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο κανόνας, ο αποστολέας, ε, καλύπτεται ως εξή. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι καλύπτονται όλες οι οντότητες ε, από τις οποίες μπορούν να προέρχονται τα παραποιημένα προϊόντα ε, το ταπεινό μου λοιπόν σχόλιο για το θέμα αυτό θα ήταν ότι δεν υπάρχει ανάγκη να... Δεν υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο. Αλλά ευχαρίστω ε, να το δούμε πιο διεξοδικά, αν πιστεύετε ότι χρειάζεται περισσότερη σαφήνεια. Αυτά έχω να σα πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τελειώσαμε με τα σημεία 4 και 5. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που έλαβαν το λόγο. Και τώρα να πάμε στο σημείο 10. non ho visto arrivare. δεν δεν τον είδα να έρχεται εδώ, αλλά τι γίνεται, δεν τον είδατε, άρα λοιπόν λειτουργεί η μέθοδος δίαιτας. Λυπάμαι, λυπάμαι που δεν είχα την ευκαιρία να ακούσω τη συνάδελφο Μπάστος, γιατί δυστυχώς δεν είμαι πανταχού παρόν δυστυχώς. Ε, ήμουν αλλού σε άλλη συνάντηση και έφτασα καθυστερημένα. Και στην προηγούμενη συνάντηση εδώ στην Επιτροπή τόνισα για αυτή τη δέσμη μέτρων για το κοινοτικό σήμα. Πρόταση που θα είναι, θα κοστίζει λιγότερα χρήματα, θα, καταγραφή σημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα βελτιώσει και τις συνθήκες για τη καινοτομία στις εταιρείες, επιχειρήσεις και την προστασία κατά των παρανομών ε, απομιμήσεων ε, εδώ. Συμφωνώ με την κυρία Μπάστος και υπέβαλα ο ίδιος τροπολογίες και θα επιμείνω κατά κάποιο τρόπο που έχουν να κάνουν ε, και με την ενίσχυση χάρη σε αυτό το σήμα και την εγγύηση όλων των νομοθεσιών σχετικά με την ελεύθερη πληροφόρηση, ενημέρωση και οι εξοδοτημένοι να μπορούν να ζητήσουν να υποβάλουν αιτήσει για να έχουν αυτά τα σήματα και να δούμε τι άλλο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη παρόλο που ξέρω ότι ποικίλουν οι απόψεις και είναι και αποκλίνουσες. Πάντως για να μπορέσουμε να έχουμε μια παρόμοια γνωμοδότηση χρειάζεται μια σύγκληση ε, από πάρα πολλές απόψεις ε, ώστε ό,τι αποφασίσουμε να έχει ισχυρό χαρακτήρα. Αυτά ήθελα να πω σχετικά με το θέμα και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο, λέει ο πρόεδρος. Πάμε παρακάτω. Η συγγήτρια, μήπως θα ήθελε κάτι να πει σε αυτό. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τον συγκεκριμένο και σαφή τρόπο με τον οποίο απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ερώτημά μου και ευχαριστώ για το άνοιγμα που για τις τροπολογίες 26, 31 κλπ. Την ανοιχτή αντιμετώπιση. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι συμμερίζομαι τα όσα είπε ο κύριος Παντσέρη προηγουμένως. Πιστεύω ότι θα πετύχουμε τελικά συνένεση που δεν είναι και επαναστατικό. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να κάνουμε μία εκτίμηση της όλης Είναι σημαντικό το θέμα για την ευρωπαϊκή οικονομία, αυτό το κοινοτικό σήμα. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε τη συνάδελφο Μπάστος. Τελειώσαμε έτσι με το τέταρτο και το πέμπτο σημείο και πάμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης για τους λογαριασμούς πληρωμών. Κλουτ, Γιούργεν Κλουτ, ο κύριος συγητής. Ενώ συντάκτρια γνωμοδότησης είναι η κυρία Γκέφχαρτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie... Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Ίσως να ξεκινήσω με ένα ευχαριστώ προς τους χειώδες εισηγητές. Τουλάχιστον ε, σε όσους, ε, όσους ε, έδωσαν σχόλια και αποδέχτηκαν ότι θα κάνουν μια δουλειά στην οποία δεν ήταν συνηθισμένη σε μορφή fast track. Που μα οδηγεί στο γεγονός ότι σήμερα ναι μεν συζητούμε την γνωμοδότησή μου, αλλά σήμερα το μεσημέρι ήδη έληξε η προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών. Και αυτό δεν οφείλεται σε μένα, αλλά στην ε, διαδικασία που επέβαλε η Επιτροπή Οικονομικών και κατ' εξαίρεση για να διευκολύνω τους συναδέλφους μου, δεν έγραψα την έκθεση στα γερμανικά, αλλά στα αγγλικά προκειμένου οι συνάδελφοι να ξέρουν τι έχω γράψει. Την αποτέχθηκαν λοιπόν οι συνάδελφοι την διαδικασία, αλλά μας διαβεβαίωσε η Επιτροπή Οικονομικών ότι στη συζήτηση για την εξέβριση βαστικών προτάσεων θα προσκληθώ στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και θα συμμετάσχω. Το επιβεβαιώνω ότι, για παράδειγμα, αύριο το πρωί έλαβα πρόσκληση προκειμένου με τον κύριο Κλούτσα και τους κοιόδης συζητητέ στην Επιτροπή Οικονομικών να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Αυτή τη διαδικασία λοιπόν ακολουθούμε σήμερα. Συμφώνησα λοιπόν να ενημερώνω διαρκώς τους κοιόδης για την διαδικασία. Από πλευρά περιεχομένου τώρα. Κατά την επεξεργασία της γνωμοδότησης, τήρησα με αυστηρότητα αυτά που αποφασίσαμε στα πλαίσια της ε, νομοθετικής πρωτοβουλίας. Δεν θα προκαλέσουν λοιπόν εκπλήξεις, έκπληξη αυτά που ε, συμπεριέλαβα στην γραμματότηση στους συναδέλφους. Σημαντικό από πολιτικής άποψης είναι το γεγονός της ενημέρωσης ε, του καταναλωτή, πάρα πολύ σημαντικό θέμα, στο οποίο έδωσε και βασική θέση και έμφαση. Θέλουμε να υπάρχει συγκρισιμότητα μεταξύ των τραπεζών σε ό,τι αφορά το άνοιγμα και τη λειτουργία, τη διαχείριση ενός τραπεζικού λογαριασμού και με την μεγαλύτερη δυνατή συγκρισιμότητα μεταξύ των τραπεζών. Ένα θέμα το οποίο είναι βασικό από άποψή μου και συζητιέται και πάρα πολύ με πολύ διστάμενες απόψεις στην ε, Επιτροπή Οικονομικών. Εγώ λοιπόν είπα ότι θεωρώ ότι θα πρέπει αυτές οι διευκολύνσεις να υπάρχουν όταν κάποιος αλλάζει τράπεζα, όχι μόνο αλλάζει μια τράπεζα σε μια άλλη τράπεζα, αλλά και από μια χώρα σε μια άλλη χώρα. Για παράδειγμα, κάποιος ο οποίος εργάζεται και πηγαίνει σε άλλη χώρα. Αυτό συνδέεται και με το θέμα του κόστους ασφαλώς, πολύ σημαντικό κεφάλαιο και αυτό και όλος ιδιαίτερος όχι μόνο με τη, σε περίπτωση μεταβίβασης λογαριασμών, αλλά και σε περίπτωση ανοίγματο λογαριασμού και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ένα βασικό λογαριασμό, όταν ανοίγει κανείς ένα βασικό λογαριασμό. Αυτό αποτελεί και τον πυρήνα της πρότασή μου και των εργασιών της Επιτροπής μας. Να διασφαλίσουμε δηλαδή ότι τα πολλά εκατομμύρια πολίτες που δεν έχουν πρόσβαση ακόμα σε τραπεζικό λογαριασμό και που επιθυμούν να έχουν τραπεζικό λογαριασμό να μπορούν πιο εύκολα να τον αποκτήσουν. Και επειδή πολλοί κόσμος ε, δεν μπορεί να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό για, λόγο, για λόγους κόστους, έχει νόημα να τους δίνετε δυνατότητα να ανοίξει ένα βασικό λογαριασμό. Με τους κανονικούς ε, όρους λειτουργίας που ισχύουν στους κανονικούς λογαριασμούς. Να μπορούν δηλαδή να πληρώνονται, να πληρώνουν το ενοικιό τους. Όλα αυτά που πλέον θεωρούνται αυτονόητα στην καθημερινή ζωή του πολίτη σήμερα. Και το σχετικό κόστος να είναι το δυνατόν χαμηλότερο, συμβολικής ε, σημασίας σε ό,τι αφορά τον βασικό αυτό λογαριασμό, προκειμένου να μην αποτελεί πρόσκομα. Και δεν μιλάμε μόνο για άτομα που δεν έχουν χρήματα, μιλάμε για εποχιακού εργάτες που βρίσκονται για κάποιες εβδομάδες σε μια χώρα, μιλάμε για νέους που σπουδάζουν ακόμα, που θέλουν να κάνουν εράσμους, πρόγραμμα ανταλλαγή και να μην αντιμετωπίζουν το πρόβλημα που συχνά αντιμετωπίζουν σε κάποιες περιπτώσεις σήμερα θέλουν να κάνουν μια σύμβαση μίσθωση σε ένα άλλο κράτο και τους λένε ότι δεν γίνεται γιατί δεν έχετε τραπεζικό λογαριασμό στη χώρα. Και στη χώρα τους λένε «Α, δεν μπορείτε να ανοίξετε λογαριασμό γιατί χρειαζόμαστε διεύθυνση για να σας ανοίξουμε λογαριασμό» και έτσι τελικά οι νέοι αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι λοιπόν ε, αυτού του είδους στην Ευρώπη που θέλουν να προσφέρω στους νέους αυτούς ανθρώπους. Αυτά είναι τα πιο βασικά σημεία. Ένα σημείο το οποίο σαφέστατα θα πρέπει να συζητήσουμε σε ό,τι αφορά τις βασικούς λογαριασμούς. Ποιες τράπεζες θα πρέπει να προσφέρουν τέτοιους βασικούς λογαριασμούς. Εγώ πιστεύω ότι για λόγους μη διακριτικής μεταχείρισης και σε ό,τι αφορά τις τράπεζες θα πρέπει όλες οι τράπεζες οι οποίες προσφέρουν ιδιωτικούς λογαριασμούς, όλες αυτές οι τράπεζες θα πρέπει να προσφέρουν και τέτοιους βασικούς λογαριασμούς. Ξέρω ότι στην Επιτροπή Οικονομικών υπάρχουν άτομα που λένε ότι φτάνει μία τράπεζα, ένα είδους τράπεζα να προσφέρει τέτοιες υπηρεσίες, αλλά θεωρώ ότι αυτό αποτελεί διακριτική μεταχείριση, ιδιαίτερος αν αυτό επιτραπεί. Γιατί αυτό θα σημαίνει κόστος για το προλογούμενο, γιατί ασφαλώς αυτό το επιπλέον κόστος που θα επιβαρύνει την τράπεζα αυτή, την εκάστοτε τράπεζα, κάπου κάπου θα πρέπει να προέλθει. Και δεν βλέπω γιατί θα πρέπει να πληρωθεί αυτό και να εξεταστούν κάποιε άλλε τράπεζε οι οποίε δεν θα υπομισθούν αυτό το επιπλέον κόστο. Αυτά είναι θέματα λοιπόν που θα πρέπει να τα συζητήσουμε. Αλλά θεωρώ ότι θα είναι και στο μέλλον καλή συνεργασία και αύριο μόλις ενημερωθώ για το προς τα που θα κινηθούν οι συμβιβαστικές προτάσεις της Επιτροπής Οικονομικών ασφαλώς και θα στραφώ προς τους εισηγητές και προς εσάς και τα κείμενα αυτά που θα λάβω θα σας τα χορηγήσω προκειμένου να έχουμε και αυτή τη βάση για τις μετέπειτα εργασίες μας. Για το χρονοδιάγραμμα δύο λόγια προκειμένου και εσείς να είστε ενήμεροι. Σήμερα λοιπόν μέχρι το μεσημέρι ε, ήταν η προθεσμία για τις τροπολογίες. 4 Νοεμβρίου θα γίνει η συζήτηση για, τη για τις συμβαστικές αυτές προτάσεις ε, που θα είναι και οι συμβαστικές προτάσεις που θα προκύψουν από την Επιτροπή Οικονομικών. Εκτός πια και αν δεν μας ικανοποιήσει καθόλου το αποτέλεσμα των συζητήσεων στην Επιτροπή Οικονομικών, στην οποία περίπτωση θα υποβάλουμε δικές μας συμβαστικές ε, τροπολογίες ή να καταδείξουμε προς τα ποια κατεύθυνση θέλουμε να κινηθούμε εμείς. Και 5 Νοεμβρίου θα γίνει η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας και θα δούμε πώς θα συνεχιστούν τα πράγματα. Σας ευχαριστώ όμως ε, και πάλι και όντες εισηγητές που αποδεχτήκατε να ακολουθήσουμε αυτό το πολύ ιδιαίτερο τρόπο εργασίας. Όπως σας είπα δεν έφταιγα εγώ. Έφταιγε η Επιτροπή Οικονομικών και κυρίως ε, η Προεδρία της Επιτροπής Οικονομικών που δεν έδειξε καμία διάθεση να δώσει παραπάνω χρόνο σε εμάς για το πολύ σημαντικό αυτό έργο μας. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Μπόρισο. Dear Mr. Chair, dear colleagues, first of all... Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρότασή της, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική κατά την εξέλιξη της ε, ενιαίας αγοράς και την ε, ε, μετακίνηση εντός της Ευρώπης όλο και περισσότερων συμπολιτών μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Γκέπχαρτ για τη δουλειά της, όπως επίσης και για όλες τις συστάσεις της. Συμφωνούμε με τις περισσότερες. Όμως ε, έχουμε μια διαφωνία όσον αφορά τον τυποποιημένο κατάλογο ονοματολογίας, ορολογίας. Πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να έχουμε έναν ε, όρο που να είναι ίδιος τουλάχιστον εντός ενός ε, κράτους μέλους, ώστε να μπορούν όλοι να έχουν ένα σημείο αναφοράς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αν δεν συμβαίνει αυτό και για λόγους συγκρισιμότητας. Επίσης, 8% ε, των πιο χρησιμοποιημένων υπηρεσιών ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να αναφέρονται, αλλά επειδή είναι διαφορετικές οι προσεγγίσεις σε κάθε χώρα, προτείνουμε 8% αλλά χωρίς να υπάρχει ένα όριο 20, χωρίς να είναι 20, γιατί σε μία περίπτωση μπορεί να είναι 25, σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να είναι 20 υπηρεσίες. Είναι επίσης πολύ καλή ιδέα να υπάρχει το switching, η μετάβαση, πάρα πολύ καλή ιδέα. Σε εθνικό επίπεδο γίνεται κάτι τέτοιο, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πάρα πολύ δοπανηρό για τις τράπεζες όταν δεν υπάρχουν αρκετές υπηρεσίες που να μπορούν να παρασχεθούν για την ώρα. Ίσως καλύτερα θα ήταν να υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα εντός, εντός ε, ε χώρα στην αρχή και μετά να περάσουμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Όσον αφορά τώρα το δικαίωμα ε, του να ανοίγει έναν λογαριασμό ε, κανείς ε, εκτός της χώρας του, Κάθε εμπορική τράπεζα θα πρέπει να είναι σε θέση να ανοίξει ένα τέτοιο είδου τραπεζικό λογαριασμό σε οποιονδήποτε θέλει. Διαφορετικά, μπορεί κανεί να ισχυριστεί ότι αυτή η τράπεζα, ε, η μοναδική τράπεζα που θα ανοίγει αυτούς τους λογαριασμούς ε, θα είναι η τράπεζα των φτωχών. Γιατί μόνο σε αυτή μπορεί να ανοίξουν το λογαριασμό τους. Αν κάθε εμπορική τράπεζα μπορεί να ανοίξει το λογαριασμό σε κάθε πελάτη, Νομίζω ότι δεν ε, υπάρχει διακριτική μεταχείριση. Επίσης πιστεύουμε ότι κάθε Ευρωπαίος πολίτης μπορεί να ανοίξει ένα λογαριασμό σε οποιαδήποτε χώρα μέλος. Αν θέλουμε να εξελίξουμε την ενιαία αγορά και εφόσον όλο και περισσότερο μετακινούμαστε και βοηθούμε έτσι την επιχειρηματικότητα, νομίζω ότι είναι χρήσιμο να μπορούν να ανοίξουν και ένα τραπεζικό λογαριασμό. Εγώ πριν από κάποια χρόνια, όταν ήμουν φοιτητή ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, άνοιξε ένα λογαριασμό, μισή μήνα μου πήρε τότε για να τον ανοίξω. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες διαδικασίες που πρέπει να τις ε, δουλέψουμε. Ίσως μπορούμε να συναντηθούμε εντός της και να συζητήσουμε τα περαιτέρω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Παρακαλώ συνάδελφε. Ο κ. Κρόιτσμαν, ε, εξ ονόματο του συναδέλφου Όλη Σμιτ, Όλη Σμιτ συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με την εισηγήτρια ότι είναι πάρα πολύ σημαντική οδηγία για την χρηματοοικονομική συμπερίληψη και την ε, ε, ομαλή κινητικότητα μακροπρόθεσμα για το on a fee σε ό,τι αφορά την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής ε, Εισηγητρίας δεν συμφωνεί. Προτιμά την προηγούμενη διατύπωση σε ό,τι αφορά ε, το μηδενικό κόστος. Συμφωνεί με την εισηγήτρια ότι αυτή η υπηρεσία θα πρέπει να μην προσφέρεται μόνο από ένα φορέα σε ό,τι αφορά τη μετάβαση, το switching. Συμφωνεί ότι θα, θα, πρέπει, να μείνει στην οδήγηση, αλλά να μην είναι δωρεάν. Και τέλος, Επίσης, ο Όλοϊ Σμιτ σε ό,τι αφορά την πληρωμή χωρίς, ε, σε, σε διάφορα νομίσματα χωρίς ε, τέλη. Δεν ξέρω να έχουν κατατεθεί σχετικές τροπολογίες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κοσνουσνίτς. Πρόεδρε, θα ήθελα τώρα να ευχαριστήσω για την σχετική προσέγγιση και θα ήθελα να υποστηρίξω την εργασία αυτή και εμείς ε, η ομάδα μας ε, θα ε, το υποστηρίξουμε αυτό για την πρόσβαση στις τράπεζες και τη συγκρισιμότητα, τη σύγκριση των ε, τιμών των τραπεζών. Δύσκολο είναι να έχει κανείς μια σταθερή σύγκριση γιατί οι τράπεζες προσπαθούν ε, να δουν τα πράγματα πως έχουν και οι τιμές δεν αποτελούν το μοναδικό παράγοντα. Ίσως θα πρέπει να προσανατολίσουμε καλύτερα τον πελάτη για αυτές τις ε, βασικές ε, συναλλαγές και κάπως ε, διστάζω όσον αφορά την πρόσβαση σε αυτό τον βασικό λογαριασμό. Χρειάζεται βέβαια να μην υπάρχει καμία διάκριση όσον αφορά τον τόπο κατοικίας ή την εθνικότητα και αυτό το να ανοίγει κανείς λογαριασμό στην τράπεζα θα πρέπει να είναι δωρεάν, αλλά στα πλαίσια αυτά δεν μπορούμε να το λύσουμε τώρα. Ευχαριστούμε. Τελευταία παρέμβαση τώρα. De Jong. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την εισηγητρία κυρία Κέπχαρτ για τη δουλειά που κάναν ένα ερώτημα σε σχέση με τη διαδικασία, γιατί άργησα λίγο. Νόμιζα στις 6 θα ξεκινήσει το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Νομίζω ότι η Επιτροπή Οίκων μας ε, έτρεξε και γι' αυτό τρέχουμε κι εμείς για την προθεσμία. Πριν την προθεσμία, προθεσμία λοιπόν υπέβαλα κάποιες τροπολογίες και υποθέτω ότι εσωτερικά θα συζητήσουμε τις τροπολογίες για να δούμε ποιοι είναι οι συμβιβασμοί από δικής μας πλευράς, ε, από πλευράς ε, οίκων. Ίνκο, συγγνώμη, όχι έκον. Θα πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε τη δική μας πορεία. Πέρα από αυτό, συμφωνώ με την εισηγήτρια σε ό,τι αφορά τις γραμμές ε, που έχει θέσει στην γνωμοδότηση. Οι τροπολογίες αφορούν λεπτομέρειες. Μία ερώτηση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα από τα θέματα τα οποία προκάλεσαν πολλές τροπολογίε είναι το εξή. Και στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην έκθεση της κυρίας Γκέπχαρτ γίνεται διαρκής αναφορά στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 για ε, κάποιες υπηρεσίες που συγκαταλέγονται στο basic payment στο βασικό αυτό λογαριασμό. Εγώ συμφωνώ ότι θα πρέπει να μιλάμε για όλες τις υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με το basic payment. Δεν τα βλέπω όμως όλα αυτά στο 5 του άρθρου 3, αλλά στην παραγράφο 2. Θα ήθελα αυτά να διαγραφούν από το 2-5, στο 5-2 δηλαδή, ε, αν ακολουθήσουμε δηλαδή τη γραμμή της κυρίας Γκέπχαρτ, το οποίο και θα ήθελα να γίνει. Και θεωρώ λοιπόν ότι από παντού και στην έκθεση Gebhardt θα πρέπει να δώσουμε σημασία να το προσέξουμε αυτό. Αν συμφωνήσουμε επί αυτό, νομίζω ότι θα γλιτώσουμε μεγάλη σύγχυση, μεγάλη φασαρία. Και αυτό που μου αρέσει στην έκθεση Gebhardt είναι ότι στο επίκεντρο είναι ο χρήστης. ένα θέμα μόνο. Αν ε, διαλέξω ένα τραπεζικό λογαριασμό, ένα πράγμα είναι το κόστος, τα χρήματα, αλλά θέλω για παράδειγμα να μην επενδύει και στην βιομηχανία όπλων, να επενδύει σε βιωσιμότητα για παράδειγμα. Αυτό τι σημαίνει ότι αν θέλουμε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια για τη τιμολόγηση, για τα τέλη, αυτό δεν σημαίνει ότι έτσι εγγυόμαστε και διαφάνεια για την πολιτική, τη στρατηγική των τραπεζών. Αναφέρεται αυτό μία φορά σε μία τροπολογία που υπέβαλα για να αναφερθεί τουλάχιστον το θέμα αυτό. Δεν αποτελεί βέβαια λύση. Θα ήθελα λοιπόν και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς την εισηγήτρια να ρωτήσω Έχετε σκεφτεί τι λύση θα μπορούσε να υπάρξει για το θέμα αυτό, γιατί ο καταναλωτής λέει ότι θέλω καλά, καλή τιμολόγηση, αλλά θέλω και μια τράπεζα που να επενδύσει στο περιβάλλον, για παράδειγμα. Μιλάμε για ποιοτικά κριτήρια, λοιπόν. Τι κάνουμε με τα κριτήρια αυτά. Ε, Σας ευχαριστώ. Η κυρία από την Επιτροπή θα μπορούσε να λάβει το λόγο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Ευχαριστώ κυρίως την κυρία Γκέπχαρτ για την πολύ καλή δουλειά της σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το εκτιμούμε ιδιαίτερο. Συμφωνώ με τον προλαλήσαντα ότι θεωρούμε ότι η έκθεση της κυρίας Γκέπχαρτ ε, ότι θέτει στο επίκεντρο τον καταναλωτή. Χαιρόμαστε πολύ και το επικροτούμε. Επίσης επικροτούμε το γεγονός ε, ότι η μετάβαση διασυνοριακά από τη μία τράπεζα στην άλλη είναι πολύ σημαντική αν θέλουμε να μιλάμε για ενία αγορά ε, οικονομικών υπηρεσιών ε, για τους καταναλωτές. Είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι ε, είναι ένα πρόβλημα πανευρωπαϊκό. Ε, δεν συμμετέχουν ε, οι καταναλωτές μας στις οικονομικές αγορές. Είναι ένα πρόβλημα. Είναι πρόβλημα όμως και για τους, για τους λογαριασμούς πληρωμών. Εμεί θελήσαμε να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Βλέπουμε το ζήτημα της προσβασιμότητας που επεκτείνεται σε πέρα από μία τράπεζα και εναγωνίως περιμένουμε ε, που θα οδηγήσουν ε, οι συζητήσεις των συνομοθετών. Εμείς τουλάχιστον ε, μία τράπεζα θα θέλαμε να ορίσουμε και μετά θα δούμε τι θα γίνει με τη συμβατότητα. Είναι πολύ δύσκολο το εγχείρημα. Προσφάτως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, οργάνωσε για τη συμπεριφορική οικονομία ε, μια διάσκεψη και ρωτήσαμε τους εμπειρογνώμονες ουσιαστικά για την ε, οικονομική εκπαίδευση. Πώς παρέχεται η οικονομική εκπαίδευση των καταναλωτών για να μπορούν να διχειριστούν όλες τις πληροφορίες που τους δίνουν οι πάροχοι λογαριασμών πληρωμών. Μπορεί να το κάνει κάποιος πολύ απλό, μπορεί να όσο και αν ε, ο άλλος εκπαιδευτεί, το σημαντικότερο τελικά είναι τι πληροφορίες θα δώσει ο κάθε φορέας. Οπότε εμείς προσπαθήσαμε να τα συμπεριλάβουμε όλα αυτά όταν πλαισιώσαμε την, πρόσταση, την πρότασή μας, να είναι τουλάχιστον σαφή τα πράγματα, να είναι σαφή η πληροφόρηση και περιεκτική. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αν ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες, αυτό δεν θα αντιβαίνει στη σαφήνεια των πληροφοριών. Αυτή είναι η μόνη πρόταση που μπορούμε να κάνουμε. Όσον αφορά τη συγκρισιμότητα, να πω ότι οι συγκριτικά εργαλεία για πρώτη φορά υπάρχουν σε νομοθετική πρόταση, γιατί έχουμε δει τέτοιου είδους πρακτική χρήση συγκριτικών εργαλείων και θέλουμε οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε τουλάχιστον ένα πρόγραμμα ε, πιστοποιημένο, ε, διαπιστευμένο. Αν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα προκειμένου να είναι αξιόπιστα ε, αυτά τα συγκριτικά εργαλεία, ευχαρίστω, αλλά πρέπει να κρατήσουμε το σύστημα σε διαχειρίσιμα επίπεδα. Η Προεδρία, η τρέχουσα Προεδρία έχει επιδείξει ιδιαίτερη πρωτοβουλία ε, οργάνωση όσο και όσο το δυνατόν περισσότερων συνεδριάσεων για να ολοκληρωθεί ανάγνωση και θα θέλαμε το Κοινοβούλιο να μας βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση για να εγκρίνουμε σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία την οδηγία αυτή. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα συμπληρώσει άλλες ε, προσπάθειες που κάνουμε για τον καταναλωτή στις δύσκολες συνθήκες μιας οικονομικής κρίσης, οπότε θα σας ε, παρέχουμε όσο ε, μπορούμε περισσότερη βοήθεια για να μπορέσουμε να το επιτύχουμε. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους και τις εισηγητές για τον πολύ επικοδομητικό τρόπο των παρεμβάσεών τους. Νομίζω, κύριε Μπόρισοφ, έχετε απόλυτο δίκιο. Θα πρέπει ασφαλώς να φροντίσουμε να χρησιμοποιούνται οι ίδιοι όροι προκειμένου να υπάρχει συνέχεια και συνέπεια. Συμφωνώ απόλυτα, λοιπόν. Το ερώτημα, λοιπόν, είναι σε ό,τι αφορά τη συγκρισιμότητα των τραπεζών εδώ θα πρέπει να το σκεφτούμε όντως. Αλλά η συγκρισιμότητα με κριτήρια που διαφέρουν από κράτος σε κράτος θεωρώ ότι δεν είναι κάτι το το εφικτό. Και σε αυτό θα πρέπει να βρούμε μια λύση λοιπόν. Εγώ θα ήθελα να υπάρχει μια γενική συγκρισιμότητα για τους πολίτες. Καταλαβαίνω φυσικά τις αντιρρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κατά πόσον αυτό θα πρέπει να γίνει σε μια συνθήκη ή όχι. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Α, α, η διάθεση των πληροφοριών, ότι θα πρέπει να διατίθενται οι πληροφορίες όταν το χρειάζονται οι πολίτες για όλες τις υπηρεσίες τις οποίες επιθυμούν να έχουν. Εδώ νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να το επιδιώξουμε αυτό. Δεν είμαι πολύ πεπισμένη κατά πόσον μιλάμε για 20%, 25%, 80%. 80% από ποιο σύνολο. Τα προϊόντα που προσφέρουν οι τράπεζες ανανεώνονται διαρκώς. Πώς υπολογίζεται λοιπόν αυτό το 80% αυτό το θέμα και το ερώτημα έθεσα κύριε Μπόρισοφ. Χρειάζομαι λοιπόν κάτι απτό για να έχω μία άποψη. Και αυτό με τα ποσοστά καλό είναι πάντα, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια σταθερή βάση. Αλλά πολύ απλά στις τραπεζικές ε, δραστηριότητες δεν υπάρχει αυτή η βάση και αυτό λοιπόν με ανησυχεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αλλαγή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό με απασχολεί ιδιαίτερως. Πριν από κάποια χρόνια ήμουν εισηγήτρια σε ό,τι αφορά τις διασυνοριακά εμβάσματα. Και το ξέρω ότι ήταν τεράστια η φασαρία που προκλήθηκε με τις τράπεζες. Ότι δεν γίνεται, είναι πολύ ακριβά αυτά, δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Δεν έχουμε τις επιχειρησιακές δυνατότητες. 100.000 λόγους προφασίστηκαν για το, για το ότι δεν μπορούσαν. Εμείς ως κοινοβούλιο επιμείναμε και σήμερα έχει περάσει. Αν δεν αυξήσουμε λοιπόν την πίεση, οτιδήποτε καινούργιο κάνουμε, ασφαλώς πάντα θα είναι αντίθετη η εμπλεκόμενη φορείς, γιατί πάντα τους κοστίζει κάτι. Το θέμα είναι, αξίζει τον κόπο, να το επιδιώξουμε, να το προσφέρουμε αυτό στους πολίτες, αυτή την ενιαία αγορά που έχουμε για τους επιχειρηματίες, να την περάσουμε και να την ε, εγγυηθούμε και για τους καταναλωτές. Και θέλω επιτέλους να κάνουμε κάτι και για τον πολίτη. Κάτι για τον καταναλωτή, όχι μόνο για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και του καθεξής. Και γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα το θέμα αυτό, με απασχολεί πάρα πολύ. Και εμένω αυτό θα το συζητήσουμε εντελεχέστερα. Σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά κριτήρια, κυρία Ντεγιόγκ, τι συμπαθητική και καλή ιδέα που είναι αυτή. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ ως τώρα, αλλά πολύ φοβάμαι ότι στο πλαίσιο του νομοθετικού αυτού πακέτου θα αποτελέσει ε, ένα υπερβολικό στοιχείο. Γιατί θα πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε υπό ποια κριτήρια θα γίνει αυτή η επιλογή θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια σχετική μελέτη. Γιατί τότε δεν θα είναι το θέμα μόνο οι τράπεζες οι οποίες δεν θα επενδύουν σε όπλα. Το θέμα είναι τι γίνεται και με τα οικολογικά κριτήρια, τα κοινωνικά κριτήρια. Υπάρχουν πάρα πολλά λοιπόν θέματα τα οποία θα έπρεπε να συμπεριληφθούν και να ληφθούν υπόψη. Ε, Βεβαίω θα ήμουν πρόθυμη να το συζητήσω το κριτήριο αυτό. Προσφάτως άλλαξα και εγώ την τράπεζά μου και ξέρω γιατί το τι μιλάω και ξέρω τι προβλήματα συνεπάγεται αυτή η αλλαγή και ασφαλώς ρώτησα την τράπεζα τι είδους επιχειρήσεις κάνει. Δεν μπόρεσαν να μου απαντήσουν. Καλό θα ήταν να μπορούσαν όμως. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν ε, μπορούμε να απορρίψουμε την ιδέα. Είναι καλή, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη φάση. Να σας υπενθυμίσω επίσης, επειδή δεν είχαν έρθει όλοι όταν το ανέφερα, να σας πω ποιο το είναι το χρονοδιάγραμμα. Αύριο το πρωί, λοιπόν, μια εισαγωγή έχω στις συμβαστικέ τροπολογίε στην Επιτροπή Οικονομικών. Θα τη συζητήσουμε, λοιπόν, από κοινού. Δεν θα τοποθετηθώ οριστικά από πλευρά τη Επιτροπή Γενικό, επειδή δεν έχω τη σχετική βάση. Θα ενημερώσω το συντομότερο δυνατόν του και συζητητέ για τι προτάσει αυτέ που θα συζητηθούν στην Επιτροπή Οικονομικών, να έχετε κι εσεί μια βάση. Και επ' αυτόν λοιπόν θα συζητήσουμε τι συμβαστικέ τροπολογίε τη Επιτροπή τη δική μα της ΕΜΚΟ. 4 Νοεμβρίου θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και στην Επιτροπή μας και η ψηφοφορία στην Επιτροπή ΙΜΚΟ προβλέπεται για 5 Νοεμβρίου. Για τις 5 Νοεμβρίου. Και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το fast track το δεχτήκαμε ακριβώς επειδή είναι σημαντικό στην τρέχουσα θετία να ολοκληρωθεί το θέμα αυτό. Ήτανε και πολιτική βούληση του Κοινοβουλίου να υποβληθεί μια τέτοια πρόταση. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να φροντίσουμε όντως να είμαστε καλά προετοιμασμένοι, αλλά να δράσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και έτσι ολοκληρώσαμε με την ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για τις ε, πραγματικά πολύ καλές τοποθετήσεις σας. Την επόμενη εβδομάδα, 5η 17 Οκτωβρίου, θα έχουμε μία συνάντηση από τις 9 μέχρι 12.30 και από τις 3 μέχρι τις 6.30 το απόγευμα. Αυτή θα είναι η επόμενή μας συνεδρίαση. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας.